Buongiorno. Se prendete posto. Καλημέρα σα, έχετε καλοσύνη να καθίσετε. Possiamo dare inizio ai lavori. È un'arma di... Allora, il primo punto all'ordine del giorno di questo... Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη για σήμερα 16. Προσβασιμότητα των ιστοτόπων των οργανισμών του δημοσίου τομέα. Με εισηγητή τον συνάδελφο Χατζημαρκάκη, στον οποίο δίνω το λόγο αμέσω και μετά περνάμε στου σκιώδει ηγητέ. Κύριε Χατζημαρκάκη, ευχαριστώ πολύ στα αγγλικά και ευχαριστώ όλου τους συναδέλφους που κατέθεσαν πολύ άριθμες τροπολογίες. Πολλές από τις οποίες πρέπει να πω 240 Μπορεί να φαίνονται πολλές, πολλές όμως είναι ταυτόσιμες μεταξύ τους. Από το πρωτότυπο κείμενο που είχε κατατεθεί σε ε, κάποια μητρική γλώσσα του συντάκτη, μέχρι τη μετάφραση άλλαξε ελαφρώς διατύπωση, αλλά στην ουσία είναι ίδιες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε πολλές δυνατότητες για συμβαστικές τροπολογίες, που δεν θα είναι πραγματικά συμβαστικές, αλλά ε, ομαδοποίηση των ε, ταυτόσημων. Θα ήθελα λοιπόν να σας εκθέσω τις προτάσεις σε κάποιους γενικούς τομείς. Υπάρχουν διαφορές, αλλά όχι τεράστιες. Σε κάποια σημεία βλέπω κάποιες μικρές διαφορές. Τα παραρτήματα καταρχάς, όπως θα θυμάστε, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει παράρτημα με τις δημόσιες υπηρεσίες που θα έπρεπε να καλύπτει η παρούσα οδηγία, μάλλον. Ωστόσο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε παράρτημα ή παραρτήματα, αλλά διάφορα επίπεδα ε, της κρατικής οργάνωσης, τα οποία θα πρέπει με τη σειρά να οργανωθούν, με πρώτες τις ε, υπηρεσίες κεντρικής κυβέρνησης και τελευταίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά τρόπον ώστε να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει παράρτημα. Η κυρία Βανιά, ωστόσο, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μας είχε προβάλει μια διαφορετική προσέγγιση και θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά. Όλοι οι σκιώδεις ηγητές, από την μια πλευρά η κυρία Βανιό από την άλλη, η οποία μάλιστα έχει υποβάλει δύο παραρτήματα. Επομένω αναμένεται αντιπαράθεση. Προθεσμίες τώρα. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ τα κράτη-μέλη και κυρίως ε, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τις πιο μικρές, οι οποίες θεωρούν ότι είναι μεγάλη η πρόκληση. Και δύσκολο έργο να καταστήσουν προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου όλες τους τις υπηρεσίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και οι όροι της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα παίξουν σημαντικό ρόλο, κυρίως στη συζήτηση με το Συμβούλιο η Λιθουανική Προεδρία ξέρουμε ότι δεν ε, κόπτεται να το βάλει στην ημερήσια της διάταξη, στην τρέχουσα Προεδρία. Θα πρέπει και εμείς λοιπόν από πλευρά μας ως Κοινοβούλιο να αντιληφθούμε και να λάβουμε υπόψη ε, αυτό το, αυτά τα δεδομένα. Εάν θέλει το Συμβούλιο να έχει ένα μέτρο το οποίο θα εισαχθεί με ταχύ τρόπο αλλά και εφικτό κατά τη διάρκεια της προσεχούς Προεδρίας Ελληνικής δηλαδή, θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτούς τους τομείς όπου υπάρχει δυνατότητα για συμβασμούς, εν προκειμένου οι ε, προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο θα έχουν κρίσιμη σημασία. Γιατί αν πιέσουμε για πολύ γρήγορες, πολύ σύντομες προθεσμίες μεταφορές, στο Συμβούλιο να μην μπορέσει να ακολουθήσει. Έχουμε λοιπόν την ε, γενική προσέγγιση, τη γενική ε, προθεσμία μάλλον, για τις περισσότερες και γενικές διατάξεις. 2014 εισαγωγή, 2016 εφαρμογή στο περιφερειακό επίπεδο, 2020 για το τοπικό, από το 2014 στην κεντρική κυβέρνηση. Ο κύριος Τρασκόφσκι, η κυρία Στάιλερ, ο κύριος Μπίλαν, Μπίλαν ε, παρουσιάζουν όμως ένα μέτωπο με μια διαφορετική και νέα προσέγγιση, όπου λένε ότι κάθε νέο περιεχόμενο που δημιουργείται με καθιονδήποτε τρόπο πρέπει απευθείας να παρουσιάζεται στον ιστότοπο. Λογικό φαίνεται αυτό. Τρεις πολιτικές ομάδες το στηρίζουν. Επομένω δεν μπορούμε να απορρίψουμε αυτή την ιδέα, θα πρέπει να την εξετάσουμε. Το παλαιότερο όμως περιεχόμενο θα πρέπει να ακολουθήσει τους όρους της μετατροπής, της μεταφοράς μάλλον, για το 2017, πράγμα το οποίο βλέπω αρκετά δύσκολο. Θα δούμε τι είδου αλλαγέ θα προκύψουν από αυτή την ε, νέα ιδέα. Ίσως στην προσεχή συνεδρία των σκιωδών στον ιστών θα πρέπει να δώσουμε πιο πολλέ λεπτομέρειε. Πάντω μου φαίνεται πολύ καλή ιδέα και προσέγγιση. Μια άλλη προσέγγιση. 16, 18, 20, τρία ορόσημα, τρεις χρονολογίες και βέβαια αυτό θα πρέπει να δούμε σε ποιο άρθρο θα εγγραφεί, αν θα πρόκειται για το άρθρο 3.2 ή για το άρθρο 10. Νομική η συζήτηση, νομοτεχνική, ε, δεν υπάρχει λόγος να την κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει το θέμα να πάει στο 3.2, ε, στην ουσία δηλαδή, στο διατακτικό. Και πάω στον τρίτο τομέα, που είναι η επέκταση του, λεπτο, της λεπτομερούς, ε, λεπτομερούς πεδίου εφαρμογής, περιεχόμενο δηλαδή των ιστοτόπων, τι θα πρέπει να έχουν, χρήσης, χρήστης και ιστότοπος. Εάν θα πρέπει ο ιστότοπος να προσφέρει και περιεχόμενο που προσφέρεται από εξωτερικούς ιστοτόπους ή όχι και τι γίνεται με την ε, παρουσίαση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. και πώς μπορούν οι σχετικές υπηρεσίες, οι ενσωματωμένες αυτές υπηρεσίες να αντιμετωπιστούν. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε εδώ συμβαστική λύση από τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι. Εκτός της τροπολογίας 97, τη σχετική με το οπτικο-ακουστικό περιεχόμενο, που μου φαίνεται δύσκολη. Δύσκολο να δεχθώ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, δηλαδή, αν ε, επιμείνουμε για την ε, περίληψη και του ακουστικού περιεχομένου. Θα είναι μεγάλες δυσκολίες η εφαρμογή αυτού του όρου, ε, όχι μόνο για τις τοπικές αρχές, αλλά και για την κεντρική κυβέρνηση. Και υπενθυμίσω ότι υπάρχουν τρία επίπεδα προσβασιμότητας στο δίκτυο. Εάν ας πούμε θέλουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, μέσω του διαδικτύου να υπάρχει προσβασιμότητα σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε εκδήλωση προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί αυτό. Ω εκ τούτου, η τροπολογία 96, Σα λέω εξ αρχή δεν βλέπω να μπαίνει σε συμβαστική πρόταση. Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών αιτήσεων επίσης, πάλι με το πρόβλημα της μετάφρασης που επεσήμανα νωρίτερα. Καλύπτεται από αρκετέ προτροπολογίε με το ίδιο νόημα. Ιστότοποι. Ανεξαρτήτως του μέσου, του μέσου που χρησιμοποιείται και της, του, ιστοτύπου, του, ιστοτόπου, του τύπου ιστοτόπου στον οποίο, από τον οποίο προσφέρεται η υπηρεσία. Η απάντηση λοιπόν θα είναι ναι ή 109, προπολογία 109, θα πρέπει να προσαρμοστεί καλύτερα στους ορισμούς του άρθρου 2. Δεν βλέπω να χρειάζεται συμβαστική εδώ. Την έχετε την αρχική πρόταση στις ε, θέσεις του ΣΥΤΕ. Πρόσθετα μέτρα. Κατάρτιση ή ε, παρουσία και επιβολή μιας, ε, ενός φορέα εποπτείας εδώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε να κάνουμε με υποχρέωση για ενθάρρυνση να αναλάβει κανείς αυτές τις, ε, να, να ενταχθεί κανείς σε αυτές τις ειδικέ διαδικασίες κατάρτισης. Πάλι αρκετά τροπολογίες του προτείνουν. Νομίζω ότι μπορούμε στο, στην ιδέα των κινήτρων να επιμείνουμε πάλι όμως χωρίς να υποχρεώνουμε κανέναν. Είναι δύσκολο, ξέρω, ίσως ε, εφαρμοστεί αυτό από τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει περισσότερο να επιμείνουμε στα κίνητρα και λιγότερο στην υποχρέωση. Συμφωνώ απολύτως με την πρόταση αυτή και βλέπω ότι μπορούμε να έχουμε συμβαστικές τροπολογίες που θα καθιστούν σαφέστερο το κείμενο. Για δε την, ε, ε, τον φορέα εποπτείας της στήρησης, Κάποιες τροπολογίες νομίζω μπορούν να ε, ενωθούν σε μία για να διευκρινιστεί καλύτερο όρος, ο ρόλος αυτού του σώματος. Και ευχαριστώ για τη συμβουλή σας. Ο προσορισμός της αρμόδιας για την εποπτεία ή ε, ε, παρακολούθηση της υλοποίησης αρχής. Υπάρχουν διάφορε προτάσεις για το πώς θα πρέπει αυτή να ορίζεται ή να διορίζεται από τα κράτη-μέλη, διάφορες διαδικασίες, τα, τα συντροπολογία 32, μηχανισμός ε, παρακολούθησης της εφαρμογής υποχρεωτικός ή μη, η υποχρέωση για συμμόρφωση στις συστάσεις του σχετικού οργανισμού από τις αρχές των κρατών μελών. Τρεις τροπολογίες προτείνουν μια διαδικασία για υποβολή προσφυγών και τις αρμοδιότητες ε, των φορέων παρακολούθησης της υλοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να τις ενώσω σε μερικές συμβαστικές, ώστε να έχουμε μια καλή λύση. Και η τελευταία, το επόμενο ερώτημα, στο σημείο υπαριθμών 6, η καταγραφή ή η δήλωση ε, εκθέσεως, υποβολή εκθέσεως Πολλοί από εσά προτείνετε μια τακτική υποβολή εκθέσεων, ετήσια ή όχι. Ίσως θα μπορούσαμε, θα το συστήσουμε μεταξύ των ε, σκιωδών. Μπορεί κάθε δύο χρόνια να, ήταν καλή, να είναι η καλή λύση ε, για να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά και τα κράτη-μέλη. Πάντως, η μύτη άλλο κάθε δύο χρόνια πρέπει να υπάρξει αυτή η υποβολή εκθέσεων, η ενημέρωση για το τι έχει συμβεί. Και το τελευταίο, που καλύπτει λίγο πολύ τους ορισμούς, και όλους τους ε, τομείς για τις συμβαστικές τροπολογίες. Επί παραδείγματι της εξουσιοδότησης. Πολύ, καλές οι ε, πολύ καλό το lobbying ορισμένων φορέων εδώ και οργανισμών και υπηρεσιών, γιατί όλες οι τροπολογίες στείλουν προς το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, η, προσαρμογή, η προσέγγιση διαφόρων συναδέλφων της Επιτροπής τίνει προς την ίδια κατεύθυνση και βέβαια δέχομαι τις τροπολογίες τους. Στον ορισμό του φορέα του, του, της υπηρεσίας δημοσίου τομέα. Έχουμε μια διαφορά μεταξύ των ομάδων. Ο κύριος Στρασκόφσκι τίνει να περιγράφει κατά ευρύτερο τρόπο τον φορέα αυτόν. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για το ε, κράτος με τη στενή του ενία, δηλαδή κεντρική κυβέρνηση και περιφέρειες, αλλά κάθε φορέα ο οποίος προσφέρει δημόσια υπηρεσία. Σε αυτό συμφωνώ και θα το συστήσουμε βεβαίως στη συνεδρία των σκιωδών οι ιστότοποι των φορέων του δημοσίου τομέα τώρα. Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να θεωρούνται ιστότοποι του δημοσίου τομέα οι φορέων του δημοσίου τομέα αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτηση. Όταν έχουμε χρηματοδότηση 5% για τον ιστότοπο που καλύπτει κάποια ζητήματα πολιτισμού Φερρυπίν που όμως δεν ανάγονται, δεν εγγράφονται στις, στα καθήκοντα της υποχρεώσης του δημοσίου εν της στενή Θα υπολογίζεται ως δημοσίου τομέα. Δεν ξέρω, ίσως μπορούμε σαν κλειδί να ορίσουμε το ποστό της χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης. Ίσως να πούμε ότι το 5% είναι πολύ χαμηλό όριο. Θα το συζητήσουμε και θα παρακαλέσω τον κύριο Τασκόφσκι που έχει καταθέσει τη σχετική τροπολογία να μου εξηγήσει στην συνέδρια των σκιωδών συγκεκριτών τι ακριβώς εννοεί και επιδιώκει. Μπορούμε νομίζω να βρούμε μια πιο συγκεκριμένη συμβαστική λύση. Τώρα το πώς θα ορίσουμε την ίδια την προσβασιμότητα ενό ιστοτόπου. και εδώ παρόμοια διατύπωση μπορεί να γίνει μια συμβιβαστική τροπολογία που να τις καλύπτει όλες τις σχετικές. Ο ορισμός του τι είναι υποβοηθητική τεχνολογία, πάλι για το χρηματοδότηση, το τι ρόλο θα παίζει η Ένωση, θα βρούμε και εκεί μια λύση. Θέμα για τα ε, κριτήρια και τους όρους της προσβασιμότητας, πάλι και εδώ θα καταθέσω μια συμβιβαστική αποδεκτή από όλους. Και τέλος μερικές τροπολογίες για την σύσταση μιας ομάδας εργασίας της Κομισιόν. Πάλι τα ίδια λένε και εδώ οι συνάδελφοι. Βλέπετε λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι θα συνεννοηθούμε με τους κοιόδης, θα κανονίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για να δούμε σε τι βαθμό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη θέση μας με εκείνη του Συμβουλίου, να συγκρίνουμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το Νοέμβριο θα τελειώσει η επεξεργασία εδώ για να υπάρξει δυνατότητα στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο να παρουσιαστεί. Αν δεν έχουμε μέχρι το Φεβρουάριο τα τελικά αποτελέσματα, τότε ο κανονισμός αυτός δεν θα εξεταστεί από αυτήν τη θητεία. Πρέπει να το δοκιμάσουμε όμως, να το προσπαθήσουμε. Θα αρχίσω συνομιλίες και με την επόμενη την ελληνική προεδρία για να τη βάλει ψηλά στην προτεραιότητε της ώστε να φαίνονται τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Γκράτσι. Ωραία. Τώρα τα σχόλια των σκιωδών Παρακαλώ όμως να περιοριστείτε να είστε σύντομοι. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε μετά την ψηφοφαρία. Η εξάλλου η συζήτηση για τις που θα γίνει άλλοτε και άλλοτε. Αρκόφσκι. Συγγνώμη πρόεδρε αλλά πρέπει σε ένα τέταρτο να φύγω. Γιατί έχω αεραπλάνο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο μετά από αυτά που άκουσα και είμαι βέβαιος ότι για τις περισσότερες τροπολογίες θα υπάρξει συμβιβασμός πόσο μάλλον που ο εισηγητής είναι πρόθυμος να συζητήσει μερικές από τις ιδέες μας. Πρέπει να συνεννοηθούμε λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο Συμβούλιο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ετοιμαστεί το θέμα όσο το δυνατόν συντομότερα γιατί αν το αφήσουμε για την επόμενη θητεία θα έχουμε παρατήσει όλες μας τις προσπάθειες. Πέντε ερωτήματα. προ οι ορισμοί. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιο ακριβώς πρέπει να είναι το περιεχόμενο όχι μόνο των ιστοτόπων αλλά και των κοινωνικών μέσων που μπορεί να χρησιμοποιούν κινητές εφαρμογές αλλά τελικά συμφωνούμε δεν υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες το, μετά το εύρος το εύρος νομίζω ότι σωστό είναι να μιλάμε για ιστοτόπους δημοσίων οργανισμών, αλλά από ό,τι είδα στους κοιόδης δεν είμαι βέβαιος ότι οι όλο και μεγαλύτεροι και μακρύτεροι κατάλογοι που στους οποίους βάζουμε τους οργανισμούς αυτούς είναι σωστή ιδέα γιατί νομίζω ότι έτσι θα τροφοδοτήσουμε, θα ενισχύσουμε όσους θέλουν να αμφισβητήσουν το χρονοδιάγραμμα αυτής της οδηγίας. Και εδώ είμαι και εγώ ανοιχτός για συμβιβασμούς. Γιατί πρέπει να βρούμε τη σωστότερη λύση για να δούμε τι θα γίνει με την οδηγία. Αυτό για το εύρος. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα χαίρομαι που αντιδράσατε θετικά στις ιδέες μας για το νέο και παλαιό περιεχόμενο. Γιατί και εγώ το σκεφτόμουν στην αρχή δεχόμουν το διαχωρισμό σας μεταξύ τοπικών και κεντρικών αρχών. Αλλά μετά κατόπιν ορίμου σκέψεως νομίζω ότι το περιεχόμενο πρέπει να διαχωρίσουμε και όχι το είδος αρχής. Και μετά για την εποπτεία και την πληροφόρηση καθώς και την επιβολή πιθανών κυρώσεων. Αυτό είναι πρόβλημα. Και εγώ ασχολούμαι με την προστασία των δεδομένων και χθες στη Βαρσοβία είχα μια σχετική διάσκεψη με οργανισμούς από όλο τον κόσμο και εταιρείε. και κάποιος από την αμερικανική πλευρά είπε ότι για τις αμερικανικές εταιρείε ο εφιάλτης είναι πώς θα εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για αυτούς μπορεί να είναι εφιάλτης αλλά για μας είναι αποτελεσματικό. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή Μπορεί να έχουμε καλή νομοθεσία, αλλά μερικά κράτη-μέλη να μην την εφαρμόζουν. Επομένως δεν πρέπει να τελειοποιήσουμε μόνο τους ορισμούς αλλά και τον τρόπο εποπτείας και εφαρμογής. Γι' αυτό μίλησα γι' αυτό το σώμα, το ειδικό σώμα για την εφαρμογή και τα μέτρα εφαρμογή, τα εφαρμοστικά μέτρα. Μετά από αυτά που είπε όμως ο εισηγητής και πάλι νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Τέλος πέμπτον, για τα τεράστια θέματα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι όπως με τη δημοκρατία που δεν είναι τέλεια αλλά κανείς δεν βρήκε τίποτα καλύτερο. Μετά μερικές τροπολογίες για τις εξαιρέσεις ως προς τις ζωντανές αναμεταδόσεις. Υπάρχουν και εδώ μερικά προβληματάκια αλλά όχι τεράστια. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι από το ΕΛΚ θα κατατεθούν πολλές τροπολογίες εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης. Καλό είναι να τις αναλύσουμε γιατί έχουν μερικές καλές ιδέες ιδιαίτερα ως προς την συνέργεια μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων αφού η δουλειά μας είναι να τελειοποιήσουμε την ενιαία αγορά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτήν φυσικά αλλά και εκτός της ενιαίας αγοράς τι συμβαίνει. Υπάρχουν και άλλες καλές ιδέες όπως τη χρησιμοποίηση πειραματικών ή πιλωτικών προγραμμάτων για πριν την εφαρμογή της οδηγίας και έπειτα εκτός από τους ανθρώπους με αναπηρίες μιλάμε και όλο πιο συχνά και για τους ηλικιωμένου. και αυτό είναι καλό επικοινωνιακός διότι πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν μιλάμε μόνο για αναπήρους αλλά για όλους και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές γιατί μερικές φορές χρησιμοποιούμε το ίντερνετ, όλοι χρησιμοποιούμε το ίντερνετ και θα έπρεπε να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εξάλλου όλοι θα μεγαλώσουμε κάποτε και πρέπει να προβλέψουμε και μέτρα για ηλικιωμένου. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το ανοιχτό σας νεύμα. Όπως σας είπα πρέπει δυστυχώς να φύγω για να πάρω ένα αεραπλάνο αλλά είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε πολύ καλά. E Τώρα για τους σοσιαλιστές Ραμόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή μας για όσα έχει κάνει για μας προσπάθησε να καταλήξει σε συμφωνία και συμβιβασμό και αξίζει τον κόπο η προσπάθεια αυτή. Βλέπω τις τροπολογίες και διαπιστώνω ότι μάλλον είναι εύκολο να υπάρξει συμβιβασμός για αυτό το σχέδιο εγγράφου που έχει τεράστια σημασία. Τρία σχόλια έχω να κάνω. Πρώτον, κάτε με, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε κάτι φιλόδοξο ως αποτέλεσμα να συμφωνήσουμε επί ενός εγγράφου και κειμένου που να τονίζει δύο πράγματα μεταξύ των τριών που θέλω να αναφέρω. Αυτά που είπε και ο συγητής. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ώστε η θέση των Ευρωβουλευτών για την οδηγία να είναι σαφής και φιλόδοξη. Γιατί πρέπει να δώσουμε κάτι, να προσφέρουμε κάτι στους χρήστες Δεύτερον, τα ίδια πλαίσια. Θα συμμετάσχουμε στις συνεδριάσεις των σκιωδών για να επιτευχθούν συμβιβασμοί τρίτων και τελευταίων. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία, να εργαστούμε γρηγορότερα, ταχύτερα, ώστε να μην παρεμποδίσουμε την έγκριση σε αυτή τη θητεία της έκθεσης. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συμφωνήσουμε στο επίπεδο της Επιτροπής μας μετά στην Ολομέλεια και γι' αυτό θα χρειαστεί ταχύτης. Ο εισηγητής ανέφερε 7 σημεία στην παρουσίασή του και νομίζω ότι περιέγραψε τέλεια το πνεύμα των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Ίσως πρέπει ακόμη να συζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα, της περιορίες κλπ. Για μένα, για μένα λέγω, το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει πρέπει να διατηρηθεί. λόγω των εμποδίων και πιέσεων που υφίστανται οι εθνικές κυβερνήσεις και οι υπηρεσίες. Αυτό το δέχομαι. Αυτό που αρνούμε όμως είναι η κατάργηση διοριών και μεταβατικών περιόδων. Χρειάζονται, χρειάζονται. Μετά για τους ορισμούς δεν υποβάλαμε τροπολογίες, μεν, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής. Δεν θα είναι και πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε και επ' αυτού. Και... Διαπιστώνω ότι πολλοί, μεταξύ των οποίων και εμείς, ζητούν αυτή τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ιδιαίτερα ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά και ορισμένες λεπτομέρειες να είναι δηλαδή λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα που μερικοί τομείς μπορεί να καλύπτονται στο εξής από την οδηγία περισσότεροι. Ούτε και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ περιοριστικό το κείμενο. Να ξέρετε λοιπόν ότι είμαστε διατεθειμένοι για συμβιβασμούς, αλλά θέλουμε να είμαστε ταυτόχρονα και φιλόδαξοι. Και γρήγοροι. Ε, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ουσιαστικά συμφωνώ με τον εισηγητή και όλους τους ε, προηγούμενους ομιλητές. Όλοι το ίδιο θέλουμε. Συμφωνούμε ότι θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής και να το καταστήσουμε πρακτικό και λειτουργικό. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα, θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε στις συζητήσεις των σχεδόν. το να επικεντρωθούμε στο περιεχόμενο είναι καλή ιδέα, γιατί είναι, εύκολα, είναι εύκολο να κάνει κανείς... Είναι πιο εύκολο μάλλον να τα κάνει κάποιος κανείς σωστά τα πράγματα από την αρχή, αντί να τα διορθώνει στη συνέχεια. Είναι λοιπόν καλή ιδέα αυτή. με τα κινητά τηλέφωνα. Σίγουρα θα πρέπει να καλύπτονται και αυτά ήδη είναι μια πολύ σημαντική πλατφόρμα και αυξάνεται συνεχώς και η σημασία τους. Επίσης, να θέλω να πω ότι πολλές φορές είναι τεχνικά πιο εύκολο να προσαρμόσει κάποιος ένα ιστότοπο ε, κινητού τηλεφώνου σε αυτή μια νέα πλατφόρμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε τον ε, όγκο των πληροφοριών και να είναι πιο ξεκάθαρη ε, η δομή. Αυτό για τι ε, εφαρμογέ στα κινητά τηλέφωνα πρέπει να γίνει έτσι και αλλιώ επειδή είναι μικρότερε οι οθόνε. Επομένω, ναι, συμφωνώ ότι σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτό το στοιχείο. Και πολλέ φορέ θα είναι και το πιο εύκολο. Ναι, όπως είπατε, πράγματι φαίνεται ότι συμφωνούμε και Είμαι σίγουρος ότι υπό την εξαιρετική ηγεσία του εισηγητή θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Ευχαριστούμε. Γέλανα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι περισσότερες παρατηρήσεις μου έχουν ήδη παρουσιαστεί σε προγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο σημαντικά για μένα θέματα και σήμερα. Διάβασα τις τροπολογίες και συμφωνώ με τις περισσότερες από αυτές. Με πολλές συμφωνώ και ελπίζω να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. 111, 112, 113 και 115 πραγματικά ταυτίζονται σχεδόν με τη δική μου 114. Χαίρομαι πολύ που αποφασίσαμε να διευρύνουμε τον αριθμό των ιστοτόπων που θα καλύπτονται από το σχέδιο οδηγία. Το ίδιο ισχύει και για αυτά τα authoring tools 115, 116, 17 και 18. Βλέπω ότι συμφωνούμε και για την 1η Ιανουαρίου 2015 για το νέο περιεχόμενο και 2017 για το παλαιό περιεχόμενο. Ωστόσο, αποφάσισα να καταθέσω τροπολογία λαμβάνοντα υπόψη ότι θα είναι δύσκολο για μένα 1η Δεκεμβρίου 2015 και 17 αντιστοίχως θα πρέπει να θέσουμε προθεσμίες. Τώρα, για την ουδετερότητα του δικτύου, είναι κάτι το οποίο ε, εντοπίζουμε στην 56 και 147 της διτροπολογίας του κ. Σακόφσκη και 84 του κ. Ραμών. Ελπίζω μαζί με τον εισηγητή να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό που να μπορέσει να υιοθετηθεί από την πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στάλερ, παρακαλώ. Ε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. 240 τροπολογίες είπατε ότι λάβατε. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι που μας απασχολεί όλους, μας ενδιαφέρει το ζήτημα και είναι πολύ χρήσιμο και αυτό να βλέπει κανείς πόσο ενδιαφέρον είναι για τους ε, συναδέλφους. Και είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση και είμαι σίγουρη ότι θα είστε επιτυχείς στην προσπάθειά σας. Είδαμε και από τις συζητήσεις ότι υπάρχει πραγματική βούληση. Αυτό που είπε και ο Ραφαέλ και περιλαμβάνεται και στην 140 τη δική μου για το νέο περιεχόμενο. Χαιρετίζουμε και τις συζητήσει με άλλους ε, και τα όσα είπαν άλλοι συνάδελφοι για το κινητό περιεχόμενο. Και τέλος, να ρωτήσω τον εισηγητή. Ανέφερε τη Λιθωνική Προεδρία, βλέπω ότι δεν είναι εδώ σήμερα, τι θεωρεί ο εισηγητής ότι θα είναι πιο χρήσιμο και ωφέλιμο για τις διαπραγματεύσει. Ο κ. Χατζημαρκάκης μιλά ελληνικά από ό,τι ξέρω, επομένω σίγουρα θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα υπό την ελληνική προεδρία. Από πλευρά εισηγητή λοιπόν, τι είναι πιο ωφέλιμο τι θα μας βοηθήσει περισσότερο να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και να φτάσουμε στις ευρωεκλογέ με μια ε, καθώς πρέπει κατάλληλη οδηγία σε ένα πιο πρακτικό πνεύμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από πλευράς Επιτροπής έχουμε τον κύριο Γιακοβίδη. Έχετε το λόγο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια παρατήρηση. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνοψίσω και εγώ τα τελευταία που ακούσαμε και εμείς βλέπουμε πόσο σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Συμφωνούμε ε, με την έκκληση του κυρίου Ραμών για ε, την ταχύτητα, για να καταφέρετε κι εσείς ε, να καταλήξετε σε συμβασμό από όσα ακούσαμε, θεωρούμε και εμείς ότι θα καταλήξετε σε συμβασμό και θα επιταχυνθεί η διαδικασία για να υπάρχουν τα απαραίτητα αποτελέσματα μέσα σε αυτή τη θητεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ορισμούς και το πεδίο εφαρμογή, θα θέλαμε πραγματικά να προσπαθήσετε να είστε τεχνικώς ορθοί. Και γι' αυτό το σκοπό είτε οι υπηρεσίε τη Επιτροπή είτε εξωτερικοί αναλυτέ μπορούν να σα βοηθήσουν. Πολλέ τροπολογίε σε τεχνικό επίπεδο είναι ασφαλμένε ή προκαλούν σύγχυση. Και θα προσπαθήσουμε να σα βοηθήσουμε. Για τα κινητά τηλέφωνα, πολλά πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οι ιστότοποι των κινητών καλύπτονται, αυτό είναι αναμφίβολο, αλλά νομίζω ότι κάποιες ε, εφαρμογές, ε, κινητά τηλέφωνα, υβριδικές εφαρμογές, ε, που βασίζονται στον ιστότοπο, η Android ή και τα δύο, δεν είναι τόσο εύκολες και δεν υπάρχει προηγούμενο ρύθμισης εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Πρέπει να σκεφτούμε και την καινοτομία, τεχνολογική πρόοδο. Επομένω, εδώ μια προσοχή απαιτείται, να μην το παρακάνουμε, αν θέλετε. Βεβαίως, πρέπει να διασφαλίσετε ότι ό,τι λέτε θα είναι ξεκάθαρο και θα στηρίζει τους ε, χρήστες, αλλά πρέπει από την άλλη να προσέξουμε να μην ξεπεράσουμε ε, και κάποια όρια με αυτόν τον κανονισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, φιλοδοξίες, ίσως είναι μάλλον υπερβολικές σε κάποια σημεία. Φέραμε και τους νομικούς μας από την Επιτροπή για να σας εξηγήσουν, αλλά δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το κείμενο της σύμβασης του ΟΗΕ, ούτε να πούμε ότι η σύμβαση του ΟΗΕ ε, τα λέει λάθος, παρότι τα ψήφισαν όλοι, εγώ θέλω να τροποποιήσω το κείμενο καλύτερα να αποφύγουμε τέτοια πράγματα. Βεβαίω είναι φιλόδοξα, ίσως θεωρείτε ότι η σύμβαση του ΟΗΕ δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη, αλλά ας το, αποφύγουμε καλύτερα. Άλλο σημείο για το πεδίο εφαρμογή. Αν δεν τροποποιήσα, αν τροποποιήσετε το 143, ιστότοπο δημόσιου φορέα, τότε δεν μπορεί κανένας να πει ε, και να επιχειρηματολογήσει για τους ιστοτόπους των ιδιωτικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα. Ας μείνουμε στο δημόσιο τομέα λοιπόν. Επίσης, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ ιστοτόπων και υπηρεσιών. Εδώ μιλούμε για ιστοτόπους, όχι υπηρεσίες που μας συνδέουν από τον έναν ιστότοπο σε άλλο και πολλές από αυτές είναι ιδιωτικές. Και αυτό προκαλεί σύγχυση. Βεβαίως χαιρετίζουμε τις νέες ιδέες για το νέο ε, και σε το παλαιό περιεχόμενο. Σίγουρα θα διευκολύνει τα πράγματα ενώ και απέναντι στο Συμβούλιο με κάποιε ιδέες ίσω θα υπάρχει καλύτερο έδαφο συμβιβασμού με το Συμβούλιο που υπάρχει αρκετή αντίδραση ε, σε ό,τι αφορά τα legacy, τι σημαίνει δηλαδή ε, αυτό το παλαιό περιεχόμενο. Είναι μια καλή προσέγγιση, όμως και πάλι θα πρέπει να υπάρξει συμβασμός μεταξύ ενός καταλόγου πολύ συγκεκριμένου και μετά ξέρουμε τι πρέπει ακριβώς να παρακολουθούμε και ε, όλων των ιστοτόπων, αλλά μετά θα πρέπει να υπάρχει ένας ρεαλιστικός μηχανισμός υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση. Επομένω, είτε θα έχουμε κατάλογο που θα είναι πιο εύκολο ε, στην παρακολούθηση και στι εκθέσει, ή παλαιό στι προθεσμίε ξεκαθαρίζει τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά πιο δύσκολο να καταλάβουμε τι παρακολουθούμε και τι ξεδιαλέγουμε. Επομένω, να δώσουμε το λόγο στον νομικό μας σύμβουλο και τον τεχνικό μας εκπρόσωπο να δώσω ακόμα μερικές εξηγήσεις. David. Δεν θα εξετάσω χωριστά κάθε τροπολογία, ωστόσο θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα, τα οποία είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. Καταρχάς ότι οι τροπολογίες δεν μπορούν να θεσπίσουν ad hoc ή επιπλέον υποχρεώσεις οι οποίες είναι συμβατε με το δευτερογενές ευρωπαϊκό ή το διεθνές δίκαιο, όπως η 83. Δεύτερον, ορισμένες τροπολογίες πρέπει να προσαρμοστούν στη νομική βάση του κειμένου, που είναι η εσωτερική αγορά. Πρέπει επίσης να γίνει σεβαστή η αρχή της αναλογικότητας. Με αυτά τα δύο όρια μπορούμε βεβαίως να συνεργαστούμε και να, κατα... να διευρύνουμε το κείμενο ώστε να γίνουν δεκτές των ατόμων τροπολογίες. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ συνάδελφοι. Ήθελα να ξεκινήσω με την Επιτροπή καταρχάς. Ήταν πολύ χρήσιμο το όταν παρούσα και στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών, τη μία που κάνουμε μέχρι τώρα, διότι υπάρχουν πολλά θέματα και νομοτεχνικά Επομένως, θα είναι καλό να είστε και στην επόμενη, ακόμη πιο κρίσιμο θα έλεγα. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις ως προς το νομοτεχνική διάσταση, αλλά Κάθριν, κύριε Μπίλαν, α, ο κύριος Στροσκοφιστικός δυστυχώς έφυγε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε όμως αγαπητοί συνάδελφοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια νέα ε, προσέγγιση, έχει δεχθεί τη νέα προσέγγιση, πρώτα το νέο περιεχόμενο και σιγά σιγά το παλαιότερο και ως εκ τούτου σας δίνω και από πλευράς μου την απάντηση και βεβαίως οι συνομιλίες με την ελληνική προεδρία θα στεφθούν με επιτυχία. Η ελληνική προεδρία χρειάζεται την επιτυχία μια ε, ένα σημείο το οποίο νομίζω μπορεί να κριθεί και πάνω σε αυτό το νομοθέτημα. Θέλουν να το παρουσιάσουν ως επιτυχία τους. Θέλουν να στεφθεί με επιτυχία για να το έχουν στο στον πίνακα αποτελεσμάτων το Ευχαριστώ πολύ. Καλά θα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες τον Οκτώβριο στην προσοχή συνεδρίαση και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Με πρώτο θέμα τη της προγράμματος δράσης για τη τελωνία και τη φορολογία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020. Παρακαλώ τον κύριο Μπαλτασάρη να μας πει αν έχει καμία δήλωση. Όχι. Δύο ψηφοφορίες πρέπει να γίνουν. Μία φορά την συμφωνία με το Συμβούλιο και η άλλη το κείμενο που θα αναγνωστεί στην αίθουσα για να ψηφιστεί και να ενσωματωθεί. Με παρακολουθείτε όλο καλό. Όχι, όχι, αυτά που σας λέει η συνάδελφος, εντάξει, συνεννοηθήκατε. Εμένα μην με υπολογίζετε. Καλώς. Λοιπόν, το κείμενο το οποίο θα πρέπει να ψηφίσουμε θα ενσωματωθεί, αφού ψηφιστεί από την ε, Ολομέλεια, στο ψήφισμα για τα τελωνία. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Το κείμενο της συμφωνίας με το Συμβούλιο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τώρα το κείμενο το οποίο θα πρέπει να αναγνωστεί στην Ολομέλεια και να ενσωματωθεί στο τελικό ψήφισμα. Άρχεται η συνεδρίαση. Η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα περνάμε. Στην ψηφοφορία για τις πρακτικές της παραπλανητικής διαφήμισης. Πρόκειται για την έκθεση του συναδέλφου De Jong. Η συμβιβαστική α παρακαλώ, υπέρ. αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Λεγκρίπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. Της κυρίας Λεγκρίπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι. Του κυρίου Πουπάκη. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να επελθέψουμε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Επτά. Πάλι γκριπ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει μόνο οκτώ. Δε γιόγκ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εννέα πουπάκι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δέκα πρέντεργαστ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έντεκα λογκρίπ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρεις τροπολογίες της κυρίας Μπέντερ Πέντεργκαστ για την αιτιολογική ε, σκέψη 12, 13 και 14 τον αριθμό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Παράγραφος 1. Κείμενο τροπολογίες της νομικής επιτροπής υπέρ. Κατά αποχές. εγκρίνονται. 15. Gris υπερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1β. 9 της Τζουρί υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 17 ροσφόρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 πάλι ροσφόρ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ας γυρίσουμε όμως πίσω γιατί ξεχάσαμε την 18 που είναι συμβατή και με την έγκριση της 17. 18 λοιπόν, Μάντερς υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε ως προσθήκη την 20 του κυρίου Χάνς Πέτερ Μάρτιν υπέρ κατά άποχες απερίφθη 21 Μάντερς υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 22 Μπίλαν υπέρ Θέλετε παλήθευση. Καλώς, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 23. Όχι, ξαναγυρνώ στην 22. Με συγχωρείτε, εμπίλαν υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 23 καταπίπτει, 24 πάλι Μπίλαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 σε δύο τμήματα. Τροπολογία που πάει εκεί. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7-2 της νομικής υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαληθεύουμε. Ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Κύριος Φόξ. Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω ότι, έχω, ότι είμαι παρόν, έχω την κάρτα μου, αλλά κανένα μηχάνημα δεν τη δέχεται. Μπορείτε τουλάχιστον να σημειώνετε αν ε, ψηφίζω δυνατά ως ισχυρό και να συμπληρώνετε στον κατάλογο τη ηλεκτρονικής ψηφοφορία. Καλώ. Παρακαλώ λοιπόν τότε και στι ηλεκτρονικέ ψηφοφορίες να σηκώνετε το χέρι για να μα δείχνετε πώ ψηφίζετε. 31. Λεγκρυπ, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 ως προσθήκη μάντες υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθη 34 μπιέλαν υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας Εγκρίνεται. 35 λεγκρίπ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 που πάει υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην 11β τώρα η 6 της τσούρ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Σαράντα πέντε υπέρ κατά απερίφθη. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 Μάρτιν Περ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 μπιέλαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρασε. Approvato all'unanimità con il voto anche del collega Fox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 Uh, Πρόεδρε, εξ ονόματος του Μάλκολμ Χάρμπορ που λείπει, αποσύρω την τροπολογία του 91. Καλά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αρχίζουμε. Τροπολογία 15 συγκητή υπέρ. Κατά. Όχι, δεν εγκρίνεται. 16 Περ, Κατά. Όχι, εγκρίνεται. Εκπίπτει η επόμενη, λοιπόν, 17 με προφορική τροποποίηση. Υπάρχει καμία αντίρρηση στην προφορική τροποποίηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Στο εξή δεν θα ρωτάω γιατί έχουμε πολλές προφορικές τροποποίησεις. Αν υπάρχει αντίρρηση να μου το λέτε πριν την ψηφοφορία για να κερδίσουμε χρόνο. 17 με την προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 του ζητητή υπέρ κατά εσ εγκρίνεται. Ci sono il 19, il 20, il 21. 19, 20, 21, 22, 23 και 24 και 25 είναι του εισηγητή με προφορικές τροποποιήσει. Προτείνω να τις ψηφίσουμε ολε μαζί. Υπέρ, επαναλαμβάνω, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 25. Λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 95 του εισηγητή πάλι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 και 96 ταυτόσημες. Σαλδελμός και d'accordo. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 97 μέντερ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 98 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Δεύτερο τμήμα. Και κοντράριο. Υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. 99 ρούλ υπέρ κατά Επαλήθωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. 100. Βάιλερ Βαντερκάμπ υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται 27 ψυχητή υπέρ κατά χες εγκρίνεται «28, 101, 102, 29 και 30 είναι όλες του εισηγητή», λέει ο Πρόεδρος. «Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί» χωρίς την 101. Καλά. Ψηφίζουμε πρώτα την 101 και μετά τις υπόλοιπες. 101 περ κατά επαλήθευση. Βοτεκίουζα. Έληξε. Ισοψηφία απορρίπτεται. Α, ναι. Α, ναι, ήσασταν κι εσείς, ναι. Αλλά πάντως απορρίπτεται. Και με την ψήφο του συναδέλφου Φόξ. 28, 102, 29, 30 υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνονται. 31, 32, 33. Μαζί υπέρ κατά ποιες εγκρίνονται 103 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 34 και 35 του εισηγητή υπέρ κατά ποιες εγκρίνονται 104 Βαντεκάμπ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 Harbor υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 και 107 ταυτόσιμες Camp και Harbor υπέρ κατά χες εγκρίνονται. 108 Harbor υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται 109 έχει καταπέσει 36 και 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 38, 39, 40, 41, 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 43, 44 και 45 υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται. 46 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 47, 48, 49, 50 και 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 110 έχει αποσυρθεί. 52 πέρ. Κατά ποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 χάρμπορ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά οχές, εγκρίνεται 56 υπέρ κατά οχές, εγκρίνεται 112 χάρμπορ υπέρ κατά επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία έληξε απορρίπτεται. Ω, όχι, όχι. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Λόγω της ψήφου του συναδέλφου μας Φώκας. Η 113 καταπίπτει, 114 επίσης, 115. Α, όχι και 115. Ωραία, 57, 58, 59, 60, Τη εισηγητρίας υπέρ κατά αποχε εγκρίνονται 61, 62, 63, 64 υπέρ και 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 66 έχει αποσύρθει 116 υπέρ κατά ελπαλήθευση. Έληξε 17 κατά με τον κύριο Φόξ, άρα απορρίπτεται. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 υπέρ κατά χες εγκρίνονται 74 και 75 υπέρ κατά χες εγκρίνονται 76-77 Κύριε Πρόεδρε τα ίδια με πριν χωρίς την 76 Ωραία πρώτα την 76 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77, 78, 79, 80, 81 υπέρ κατά εσ εγκρίνονται. 82, 83, 84 υπέρ κατά χες εγκρίνονται. 85 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 117 Βάιλερ και Βαντεκάμπ υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται. Μια στιγμή τώρα να δω. Ναι, 88 Βάιλερ υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται. Κατά πίπτη 1 ή 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 προφορική σαλτεμόζη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 αποσύρεται, 92. Βάιλερ Βαντεκάμπ. Με προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 5 καταπίπτει, 91 αποσύρεται. υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται Επτά υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται Η 93 έχει αποσύρθει, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14. 8, 9, 10, 11, 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 13 υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Έχουν αποσυρθεί 120 και 118, 119. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86. της εισηγητρίας κυρίας Βάιλερ με προφορική τροπή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 έχει αποσυρθεί. 122. Χάρμπορ, προφορική τροποποίηση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123. Βαντεκάμπ, πέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνολική ψηφοφορία για την έκθεση άρχεται ηλεκτρονικά. Έλξε. ...35 με τον κύριο Φόξ υπέρ, καμία ψήφος κατά, ούτε αποχή, ομόφωνη έγκριση, συγχαρητήρια. Ας επιστρέψουμε τώρα στη συζήτηση. Αν έχετε την καλοσύνη, αποχωρήστε ήσυχα. για να μην ενοχλήσουμε όσους θέλουν να τον λόγο. Κυρία, κυρία Χάντσλικ, φαίνεται απίθαρχη σήμερα. Ah. Bene. Ciao. Λοιπόν, το επόμενο σημείο στην μέσα διάταξη είναι το 20. Για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάγερ. που είναι εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία χρόνια, 34% όλων των πτήσεων στη Γερμανία είχαν καθυστέρηση είναι πολύ δύσκολο να διαμαρτυρηθεί κάποιος ε, ε, και να εισακουστούν ε, οι παρατηρήσεις του ή τα παραπονά του. Πολλές φορές, ακόμα και επιβάτες που έχουν πραγματικά παράπονα για τις καθυστερήσεις τις πολύ λίγες φορές παίρνουν αποζημίωση, ελάχιστο ποσοστό. Εδώ μιλούμε για τα δικαιώματα των επιβατών, όχι τα δικαιώματα των αεροπορικών εταιριών. Γι' αυτό και ο στόχο μας δεν θα πρέπει να είναι να καταστρέψουμε τις αεροπορικές, αυτό είναι αυτονόητο. Όμως, στόχος μας θα πρέπει να είναι να ενθαρρύνουμε τις αεροπορικές να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Το 34% των πτήσεων να έχει καθυστέρηση δεν είναι μια αποδεκτή κατάσταση. Όταν ο επιβάτης ε, αγοράζει ένα εισιτήριο, μπαίνει σε μια σύμβαση, ε, σε μια συμβατική συμφωνία με την ε, εταιρεία και αυτή η σύμβαση δεν μπορεί να καταργηθεί μονομερώς χωρίς να υπάρξει απαραίτητη αποζημίωση. Εγώ έχω επιφέρει κάποιες αλλαγές στην έκθεσή μου που θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα. Πρώτον, η Επιτροπή θέλει να υπάρχει κατηγοριοποίηση 5, 9 και 12 ωρών. Μια τριχοτόμηση. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει διχοτόμηση. Δύο κατηγορίες δηλαδή, δύο ώρες που θα επιφέρει ένα επίπεδο αποζημίωσης και μετά υπάρχει και ένα όριο χιλιομετρικό. Και στη δεύτερη κατηγορία, πάνω από τα 3.500 χιλιόμετρα ή πάνω από 5 ώρες καθυστέρηση. Και τότε θα έχουμε 600 ευρώ αποζημίωση και όχι 250 που είναι στην πρώτη κατηγορία. Βασιζόμαστε στην αρχή ότι η αρχική τιμή θα επιδέχεται ενός συγκεκριμένου ορίου προσάξησης. Τώρα, στην πτήση, αν υπάρχει καθυστέρηση και στις δύο πτήσεις, βεβαίως θα υπάρξει διπλή αποζημίωση, αλλά θα υπάρχει ένα όριο ανά ε, εισιτήριο, που είναι αυτό το όριο των 600 ευρώ που έχω θέσει. Βεβαίως, η ευθύνη μιας εταιρείας θα πρέπει να συνδέεται και με ε, την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, ο χρήστης. Δεν είναι δυνατόν ε, ο επιβάτης να πρέπει να περιμένει δύο ώρες όταν υπάρχει καθυστέρηση πριν έχει πρόσβεση σε δικαιώματα όπως η παροχή νερού ε, ή φαγητού. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν. και τα ίδια τα αεροδρόμια, οι θα πρέπει να υποχρεούνται να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο εάν οι αερογραμμές δεν ε, πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, νερό και ένα μικρό γεύμα είναι απαραίτητα στο πλαίσιο της ε, παροχής υπηρεσίας. Υπάρχει ένα όριο δύο ωρών. Αν περάσουν οι δύο ώρες αναμονής, ο επιβάτης θα πρέπει να δικαιούται να λάβει κάτι. Δεύτερον, ο χρόνος αναμονή για τις αποσκευές δεν ρυθμίζεται αυτή τη στιγμή, όμως προτείνουμε δύο ώρες. Η Επιτροπή προτείνει πέντε ώρες. Φανταστείτε τώρα να έχετε μία ώρα καθυστέρηση στην πτήση και μετά να πρέπει να περιμένετε για άλλε δύο ώρε για να πάρετε τις αποσκευές σας. Οι πέντε ώρες που προτείνει η Επιτροπή λοιπόν είναι υπερβολικός χρόνος. Άλλες διατάξεις θα πρέπει να ε, αρχίσουν να ισχύουν μετά από το όριο των τριών ε, ωρών στην καθυστέρηση. 12 ώρες έχει θέσει η Επιτροπή. Ε, είναι πολύ ευρύ αυτό το χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο είναι δυνατόν να εξισορροπήσουμε καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αερογραμμών και επιβατών. Όταν μια αεροπορική εταιρεία ανακοινώνει ότι δεν μπορεί να ε, εκπληρώσει την, ε, ε, πραγματοποιήσει την πτήση μέσα στο επόμενο τρίωρο και θέλει και άλλες ώρες, τότε υπάρχει πρόβλημα. Στην περίπτωση ακύρωσης η Επιτροπή λέει ότι ε, θα πληρώνεται, θα καταβάλει τον τίτυπο της ε, διαμονής για τρεις νύχτες. Όμως δεν φτάνει αυτό για μας. Εάν ο ίδιος επιβάτης θα πρέπει να ψάξει για διαμονή, ε, μπορεί αυτό να αποβεί ιδιαίτερα κοστοβόρο. Επομένως προτείνουμε αύξηση στα 150 ευρώ ανανύχτα. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε Άλλοι συνάδελφοι θα προτείνουν κάτι διαφορετικό. Όμως πάντα γίνεται αυτή η αναφορά στις ε, αεροπορικές, οι οποίες μπορούν να ε, κάνουν κρατήσεις ε, σε ξενοδοχεία, σε περίπτωση καθυστερήσεων ή ακυρώσεων. Και εκείνοι να πληρώσουν λιγότερα για την ίδια τιμή του δωματίου. Τώρα, το επόμενο σύνολο που θέλω να αναφέρω. Στο σύνολο ε, του φακέλου χρειαζόμαστε πιο ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα με προθεσμίες. Στόχος είναι να διευκρινίσουμε ε, οποιαδήποτε σημεία σύγχυσης. Θέλουμε να αποζημιώσουμε τους επιβάτες ε, για νομότυπα παράπονα. Θέλετε, θα πρέπει να υπάρξει μια ασφάλεια υπηρεσιών εδώ με επικαιροποίηση ετησίως των ε, στοιχείων που διαθέτουμε. Αυτό έχει ήδη θεσμοθετηθεί ε, στο Ευρωπαϊκό Χρονιστικό Πλαίσιο. Υπάρχει ήδη διετής προθεσμία. Τώρα, σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις ε, στην πρόταση της Επιτροπής οι ίδιοι επιβάτες θα πρέπει να αναλάβουν ε, το κόστος ε, των καθυστερήσεων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση απεργίας θεωρείται ε, περίπτωση υπεράνω βίας. Όμως δεν ξέρω αν ισχύει αυτό όταν είναι εσωτερικά μέσα στην εταιρεία. Αν το προσωπικό της εταιρείας απεργεί, τότε αυτό δεν αφορά όλες τις εταιρείες. Η ίδια εταιρεία λοιπόν θα πρέπει να απομειστεί το βάρος. Επίσης, θα πρέπει να καταστεί πιο ξεκάθαρο αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες και αυτό οδήγησε στην καθυστέρηση, αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε πλήρως και να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει την περίπτωση. Αποζημίωση και άλλες προβλέψεις θα πρέπει να υπάρχουν και για ε, τις περιπτώσεις Ε, όπου η πτήση αναχωρεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να ενημερώσει τους επιβάτες αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άλλο σημείο. Υπάρχει υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για επιπρόσθετες, ε, επιπρόσθετα αιτήματα αποζημίωσης. Η Επιτροπή δεν το ανέφερε στην ε, πρότασή της. Εγώ κατέθεσα τροπολογία όπου αναφέρεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διακανονισμός σε περίπτωση αποζημίωσης ή αίτησης αποζημίωσης. Κάθε επιβάτης, επομένως, που δικαιούται αίτημα αποζημίωσης ε, θα πρέπει να έχει την απαραίτητη αποζημίωση. Δεν μπορεί να υπάρξει, λοιπόν, μεμονωμένη διαπραγμάτευση με ε, κάθε επιβάτη. Αν υπάρχουν επιπρόσθετες λοιπόν ε, αιτήματα για αποζημίωση, δεν μπορεί να γίνει αυτό μεμονωμένα ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους επιβάτες. Άλλο σημείο καθοριστικής σημασίας είναι αυτό που εισήγαγα εγώ για τις ε, επιπρόσθετες ε, κυρώσεις. Υπάρχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όμως αυτό δεν φτάνει οι αεροπορικές εταιρείε θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να δίνουν τις σωστές, τις κατάλληλες πληροφορίες γιατί καθυστέρησε ή ε, ακυρώθηκε μια πτήση. Και ξέρουμε ότι πολλές φορές δεν λαμβάνουμε τέτοια πληροφόρηση. Στην έκθεσή μου λέω ότι θα πρέπει να ε, θεσμοθετηθούν κυρώσεις όταν δεν δίνονται πληροφορίες ή δίνονται ψευδείς πληροφορίες. Γιατί για να έχει ο επιβάτης πρόσβαση στα νόμιμα του δικαιώματα, θα πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησης της ακύρωσης. Επομένως, πληροφορίες ε, που δίνονται από την αεροπορική ε, στους επιβάτες πρέπει να είναι σωστές. Μετά, προσβασιμότητα της ε, κατάθεσης παραπώνων, της υποβολής παραπώνων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία, το έχουμε ήδη συζητήσει και σε άλλα πεδία είναι προς όφελος των ε, καταναλωτών και πάλι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα κατάλληλα σημεία επαφής για να διευκρινιστεί αν ε, η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη ή όχι. Ε, επαρκεί η προθεσμία των 90 ημερών για την επεξεργασία του αιτήματο. Φτάνουν 90 ημέρες. Όταν δεν τηρείται αυτή η προθεσμία των 90 ημερών, δεν δίδεται δηλαδή απάντηση, τότε θα πρέπει να έχουμε επιπλέον διατάξεις. Γιατί η προθεσμία των τριών μηνών για να λάβει κάποιε πληροφορίες για μια πτήση, προφανώς και επαρκεί. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω που είναι σημαντικό. Οι αεροπορικές γραμμές πολλές φορές λένε ότι ε, όταν η πτήση δεν είναι αρκετά επικερδής για μας, τότε απλώς ακυρώνουμε. Αυτό αναφέρεται στα, μικρά, στα ψηλά γράμματα ε, στο συμβόλαιο. Αυτό είναι μια πραγματικά αδικαιολόγητη απειλή εκ μέρους των αεροπορικών εταιριών. Αυτά ήταν τα κύρια σημεία που ήθελα να φέρω. Υπάρχουν 92 τροπολογίες και σίγουρα θα προσταθούν μία-δύο εκ μέρους μου. Προσβλέπω ε, στις ε, συνομιλίες με τους ε, συναδέλφους. Θέλω να ακούσω κριτικές παρατηρήσεις και Συμπερασματικά, ο εισηγητής της Επιτροπής Μεταφορών θα πάρει τώρα το λόγο και ε, θα τα συζητήσουμε και μαζί του για να υπάρξει και μια ε, συζήτηση μεταξύ επιτροπών. Ευχαριστώ. Α, σας ευχαριστώ. Θα δώσω αμέσως λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπακ που είναι εισηγητής ε, για την Επιτροπή, Συντάξεων Ομοδότηση, μάλλον για την Επιτροπή μεταφορά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω εδώ. Για να, περάσω, για να εξηγήσω τις ε, θέσεις μου. Βασικά στάθηκα πάνω σε τρία στοιχεία, έλαβα υπόψη βέβαια και ανέλησα τις ε, πολυάριθμες δικαστικές αποφάσεις. Δεύτερον, θεωρώ ότι όταν υπάρχει, όταν υπάρχει σύναψη συμβάσεως πρέπει να τηρείται αυτή για τα δύο μέρη. Και δεύτερον, τρίτον, πρέπει να επιδιωχθεί η ενίσχυση, η εφαρμογή και η επιβολή της ενίσχυσης των, των δικαιωμάτων του πελάτη. Ο επιβάτης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πελάτης πάντα και να μην επιδεινώνεται η κατάσταση εις βάρος του. Πολλά σημεία βλέπω να μας βρίσκουν σύμφωνους, ε, επί παραδείγματι η υποχρέωση για αποζημίωση ύστερα από καθυστερήσεις τριών ωρών στις ευρωπαϊκές και πέντε ωρών στις διεθνείς πτήσεις, η πρόταση της Επιτροπής επιδεινώνει την κατάσταση, όπως αυτή ισχύει τώρα, η, διαμά... διαβάθμιση του κυρίου Μάιερ, διπλή αυτή η διαβάθμιση δύο και τριών ώρων, επίσης αντικατοπλίστηκε στη δική μου γνωμοδότηση. Άλλα σημεία συμφωνίας σε σχέση με την δυνατότητα εξόδου από το αεροπλάνο. Δεν μπορεί κανείς υποχρεωθεί να περιμένει πέντε ώρες για να βγει από το αεροπλάνο. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό της διαφάνειας και της υποχρεώσης για ενημέρωση. Όταν κάτι όχι απλώς έχει πάει στραβά, αλλά και εκ των προτέρων, όταν υπάρχουν δεδομένα κατά την κράτηση ή κατά την ε, επιβίβαση, ε, εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο, κάποια πληροφορία, πρέπει αυτή να διατίθεται στον επιβάτη, παύλα, πελάτη, στο κάθε αεροδρόμιο, έτσι ώστε να γνωρίζει καλά πώς ε, και σε ποιον μπορεί να απευθυνθεί, θα, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την υπηρεσία στην οποία μπορεί, μπορεί κανείς να αποτανθεί. Ένα άλλο θέμα, οι άκρος εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να διευκρινιστούν πολύ πιο προσεκτικά και συγκεκριμένα γιατί μπορούν να αποτελέσουν μια, ε, ένα πρόσχημα ε, που επικαλούνται οι αεροπορικές εταιρείε για να αποφύγουν την καταβολή των αποζημιώσεων. Το ζήτημα δε των αποσκευών. Πάλι διαφορετικές μέθοδοι υπάρχουν ώστε να ε, αντιμετωπιστεί αυτή η ε, μονολυθική προσέγγιση, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ ευρύτερη διατύπωση. Ένα πρόσθετο σημείο σχετικό με την ε, πτώχευση μιας εταιρείας το οποίο βλέπω να αντιμετωπίσετε με περιθωριακό μόνο τρόπο. Δεν μπορούμε όμως να το αγνοήσουμε, γιατί ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσεως ενδέχεται το φαινόμενο αυτό να ενταθεί. Και ιδιαίτερα στις καταποκοπήν, στα καταποκοπήν οργανωμένα ταξίδια ε, μπορεί αυτό να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον επιβάτη. Ιδιαίτερα την ώρα λοιπόν που εμφανίζεται πρόβλημα ε, ρευστότητας ή και πτώχευση της εταιρεία πρέπει να μπορεί να προστατεύεται ο επιβάτης. Μια πρόταση του κύριου Μάιερ που εγώ δεν δέχομαι είναι αυτή της αναλογικότητας της αποζημίωσης ως προς την τιμή του εισιτηρίου. Φυσικά θα υπάρχουν και ε, επιχειρήματα τα οποία υποστηρίζουν αυτή την επιλογή της αναλογικότητας δηλαδή, αλλά εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που πρώτο συντάχθηκε αυτή η νομοθεσία, ο νομοθέτης είχε επιλέξει την ενιαία αποζημίωση και όχι την αναλογικότητα. Εξάλλου η αναλογικότητα θα πρέπει να ε, σημάνει αρκετά περίπλοκους υπολογισμούς και για την αξία και τα συνολικά ποσά, αλλά ενδεχομένως να οδηγήσει και σε νομικά προβλήματα. γιατί το να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες ζημίες, ένα σημαντικό ραντεβού ή κάποια άλλη πτήση που ενδεχομένω χάνει κανείς, θα μας περιπλέξει πάρα πολύ την εικόνα και εκεί πέρα βέβαια πέφτουν, μπαίνουν και άλλα ζητήματα και διεθνών συμβάσεων. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία και εμείς από την Επιτροπή των Μεταφορών θα συζητήσουμε ασφαλώς μαζί με τον εισηγητή σας βεβαίως πιστεύω ότι θα έχω αρκετές ακόμα συναντήσεις ώστε να συζητήσουμε το θέμα αυτό λεπτομερώς και να καταθέσουμε μια καλή πρόταση νομοθετική προς το συμφέρον του επιβάτη. Σας ευχαριστώ για την επικοδομητική αυτή στάση. Τώρα θα ακούσουμε τους σκιώδεις. Κυρία Βέστφαλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μάιερ, σήμερα κάναμε ένα πρωινό εργασίας μαζί. Και με τον κύριο Μπαχ βεβαίως και εμείς από την ΙΜΚΟ παρουσιάσαμε ένα πολύ καλό κείμενο πιστεύω που προστατεύει τον καταναλωτή και που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για βελτίωση αυτής της προστασίας. Όντως κύριε Μάιερ η πρότασή σας εξασφαλίζει για τον καταναλωτή, άνδρα ή γυναίκα, πολύ καλύτερη προστασία και εξασφάλιση των δικαιωμάτων του. Και βεβαίως αυτό θα κριθεί και από την δυνατότητα μεταφοράς στην πράξη αυτής της νομοθεσίας. Πώ δηλαδή μπορούμε σε καθυστερήσει σε αεροδρόμια, σε, από αεροπορικέ εταιρείε κτλ. να επιβάλλουμε αυτή την, την τήρηση αυτών των διατάξεων. Αυτό νομίζω που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ζήσει και οι ίδιοι τόσες πολλές φορές. Θα το συζητήσαμε ήδη την Δευτέρα. Ε, πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν, πιστεύω, και οφείλουν να αλλάξουν από την πρόσθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να ε, επαληθευτεί το ζήτημα των εκτάκτων περιστάσεων και να οριστεί ένας εξαντλητικός κατάλογος, να μην έχουμε δηλαδή απεριόριστη διεύρυνση αυτού του ε, όρου. Και λόγος, βέβαια θα πρέπει να παρακολουθούμε πόσο οι αεροπορικές εταιρείες η κάθε μία χειρίζεται το θέμα αυτό. Ναι, μέλημά μας είναι η διεύρυνση και βελτίωση βέβαια της ε, γνωμοδότησής σας. Έχουμε σε πολλούς τομείς σύμπτωση απόψεων. Μέλημά μας κοινό είναι η προστασία του καταναλωτή και πιστεύω ότι μπορούμε να ε, ετοιμάσουμε και να εγκρίνουμε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Άλντε, Ροσφόχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα αρχίσω με ένα αστιακή. Οι υπάλληλοι και συνάδελφοι βουλευτές εκπώνησαν ένα εξαίρετο κείμενο, αλλά ε, για να είμαστε γιατί είναι βέβαια ευφιέστατοι, αλλά και για να μην γελιόμαστε, γιατί τα έχουμε ζήσει οι ίδιοι. Ποιος δεν έχει αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίε τόσες φορές στη ζωή του. Έχουμε λοιπόν προσωπική μαρτυρία να προσφέρουμε στην υπόθεση αυτή. Άρα καλό είναι όταν μιλάμε για πράγματα που γνωρίζουμε ε, από προσωπική εμπειρία. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί το θετικό δίκαιο αφενός, με βελτίωση των δικαιωμάτων του καταναλωτή και εδώ πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι προτάσεις των, ε, του εισηγητού είναι πολύ καλές και ευστοχές ταυτόχρονα θα πρέπει να βελτιώσουμε και το, ε, την πρακτική όψη, δηλαδή τις ε, διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες και τις συνέπειες αυτών των ταλαιπωριών που υφίσταται ο Έχουμε συστήσει λοιπόν το θετικό δίκαιο, αλλά μην ξεχνάμε και τον τρόπο εξάσκησης του δικαιώματος του ε, επιβάτη. Ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων. και θα έλεγα ότι καλό θα είναι να μην χαθούμε μεταξύ των ε, θεμάτων που αφορούν διάρκεια, ποσά και ούτω καθεξής, πιο μεγάλη διάρκεια, πιο μικρό ποσό. Δεν είμαστε και ειδικοί, ασφαλώς θα πρέπει να ακούσουμε τη, τη γνώμη εκείνων που κατέχουν καλύτερα τα πράγματα. Παράδειγμα, σημαντική καθυστέρηση λόγω ενέργειας κυκλοφορίας και πρόταση από τον εισηγητή για περικοπή της ε, περίοδου των 12 ωρών σε 3 ώρες όταν ο αερομεταφορέας έχει υπετιότητα. Δεν είναι πολύ σύντομο αυτό. Χωρίς να έχω εργαστεί εγώ στον χώρο των αερομεταφορών και της αεροπορίας, αλλά επειδή έχω συζητήσει με, αρχι... αρκετούς από τους ειδικούς, ε, ξέρω ότι επικρατεί η θεωρία των ντόμινο. Όταν δηλαδή κάτι πάει στραβά σε μία πτήση, ακολουθούν προβλήματα σε όλες τις ακόλουθες πτήσεις. Αν αρχίσει ένα αεροπλάνο, τότε παρουσιάζονται καθυστερήσεις διαδοχικές ε, και στις υπόλοιπες πτήσεις. Επομένως, καλό θα ήταν να μην... Ε, να μην προκαλέσουμε ασφυξία στην ίδια την αεροπορική εταιρεία από κάτι από ένα μέτρο υπερβολικά ακραίο. Άλλο βέβαια υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό, τα αεροπλάνα κτλ. Ε, σωστό θα ήταν να βρούμε μια χρυσή τομή, ίσως το οι 12 ώρες να ήταν υπερβολική, ε, ε, υπερβολικά χαλαρές, οι 3 ώρες ίσως είναι υπερβολικά στενή προθεσμία για να αναλάβει την ε, σχετική δράση για αναμεταβίβαση εταιρεία, ε, ίσως να βρούμε κάπου αλλού την χρυσή τομή. Επίσης για την επιβολή ενός ε, παγίου ποσού ανταπόδοσης ή αποζημίωσης ή αναλογικού. Ασφαλώς καλό είναι να υπάρχει ένα πάγιο ποσό, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να λησμονούμε και το, ε, την έννοια ότι η αναλογική αποζημίωση θα πρέπει να είναι ικανοποιητική για τον, ε, προσφέρει μάλλον μια ικανοποιητική για τον επιβάτη λύση. Για δε την πίστα, το τάρμακ. όταν πια έχει αρχίσει να τροχιοδρομεί το αεροπλάνο ή μάλλον καλύτερα όταν έχουν επιβαστεί στο αεροπλάνο οι επιβάτες. Πόσες φορές δεν έχει πει ο κυβερνήτης, ξέρω ότι έχουμε μείνει μέσα στο αεροπλάνο κολλημένοι 4 ώρες, 5 ώρες και δεν έχουμε αρχίσει να τροχιοδρομούμε, αλλά αν τώρα αποβιβαστείτε χάνουμε τη σειρά μας για την απογείωση. Άρα υπάρχει επιλογή μεν της απο, αποβίβασης, μεν όλων των επιβατών, το αεροπλάνο όμω χάνει τη σειρά του, στη σειρά, στην ουρά των αεροπλάνων για αποβίβαση και μπαίνει τελευταίο. Άρα περισσότερες ακόμα καθυστερήσεις. Και μην λησμονούμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε και να ενσωματώσουμε σε όλη αυτή την ιστορία και τι ευθύνε των αεροδρομίων. Και φυσικά κάνοντα μια διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών αεροδρομίων, γιατί τα μικρά δεν έχουν τη δυνατότητα αντίδραση σε κάποιο πρόβλημα που ενδεχομένω εμφανίζεται. Αλλά υπάρχουν οι φορεί, συμβατικοί φορεί, η αεροπορική εταιρεία με την οποία συμβάλλομαι, αλλά και άλλοι ε, έξω συμβατικοί φορεί αεροδρόμια, εν προκειμένου μεγάλα αεροδρόμια, των οποίο ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Υποστηρίζω λοιπόν ε, την ε, ε, πρόταση για την αντιμετώπιση των όλων ιδιαίτερων συνθήκων του εισηγητή και της ανώτατη, του περιορισμού σε δύο το πολύ νύχτες και 150 ευρώ για το ξενοδοχείο γιατί βέβαια τα 100 ευρώ δεν αρκούσαν για την αποζημίωση της εκτέρευσης. Εν γέννη νομίζω μπορούμε να πούμε ότι βρίσκει μια καλή ισορροπία η έκθεση. Η έννοια ενός καταλόγου μη εξαντλητικού νομίζω ότι είναι καλή ε, για το τι σημαίνει έκτακτες περιστάσεις, γιατί μπορεί σήμερα κάτι που θεωρείται έκτακτη περίσταση να μην πρέπει να θεωρείται και στο μέλλον, όπως πολύ σωστά λέει ο εισηγητής. Επίση, η ιδέα της ε, διαβάθμισης ή ε, της κατάρτισης ενός καταλόγου με σειρά προτεραιότητας ή σημασία των εξαιρετικών περιστάσεων. Κοιτάξτε, εάν κάνουμε έναν κατάλογο των περιστάσεων που δεν μπορούν, αρνητικό δηλαδή, εκείνων που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ε, έκτακτες, τότε δεν χρειάζεται να γίνει διαβάθμιση και να οριστεί σειρά προτεραιότητας. αδίποτε από αυτέ τι περιστάσει δεν θα μπορεί να επικληθεί ω έκτακτη. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υποχρέωση για χορήγηση συστηματικά πληροφόρησης 30, στον επιβάτη 30 λεπτά εφόσον παρέλθουν 30 λεπτά από την οριστήσα ώρα αποχώρησης ή απογείωσης. Ε, ο εισηγητής λέει 30 λεπτά πριν. Εγώ κεντρός, ξέρω θα μου πείτε ότι είμαι όπως πάντα, αλλά το δέχομαι. Ε, θα έλεγα την ώρα της απογείωσης. Εάν δεν υπάρχει, αν δεν έγκυρη απογείωση, να ενημερώνετε τότε ο, εισηγητή, ο επιβάτης. Πάντως υπάρχουν πολλές καλές προτάσεις όπως είπαμε. Στο θέμα των ε, αποσκευών και δι των χείρα αποσκευών θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να βρούμε λύσεις ε, κατανοητές και αποδεκτές για τον επιβάτη. Ε, και επίσης μην ξεχνάμε και το σύστημα του duty free. Όταν κάνει κανείς τα ψώνια του στο duty free του αεροδρομίου Καταλογίζεται αυτό στην ε, χειραποσκευή ή θεωρείται μια επιπλέον χειραποσκευή, γιατί πολλοί ε, βρέθηκαν ενώπιον της δυσάρεσης εκπλήσεως αφού είχαν δώσει τις ε, αποσκευές τους να χρεωθούν με επιπλέον χειραποσκευή γιατί είχαν αγοράσει ένα μπουκάλι ουίσκι στο duty free του αεροδρομίου. Και ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό του non-show, της μη εμφάνισης επιβάτη. Δεν μπορεί να απαγορεύει δηλαδή η εταιρεία την επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για κάποιον ο οποίος, ε, και για τον μόνο λόγο ότι κάποιος δεν πήρε την πτήση του πήγαινε. Ξέρετε ότι αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή για τις αεροπορικές εταιρείες, είναι ένα ζήτημα το οποίο θεωρούν ότι ανήκει στα εμπορικά τους πακέτα κτλ. Αλλά πολλές φορές δεν επιλέγει ο επιβάτης ο ίδιος να μην παρουσιαστεί σε μια πτήση στο πήγαινε. Στη δε επιστροφή θέλει να επιβιβαστεί. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να αποτελέσει λόγο άρνησης επιβίβασης για τον αερομεταφορέα, τον on-show στο πήγαινε. Από την άλλη, όταν αερομεταφορέας ε, πολλά, πολύ ένα ε, αλέ ή ρετούρ ανεξαρτήτως, το οποίο όμως έχει πολλές μεταπιβιβάσεις και συν, συνδυασμένες πτήσεις, τότε προφανώς θα πρέπει και ο επιβάτης να τηρήσει αυτή την σειρά Εάν έχει ένα κυκλικό εισιτήριο και χάσει την μία από τις πτήσεις της, από την πρώτη πτήση, δεν μπορεί να εμφανιστεί στην επόμενη μεθεπόμενη πτήση, γιατί αυτό θα σήμαινε βέβαια απόλυτη ανταγωνιστικότητα ως προς τις ε, τιμολογιακές προτάσεις, ε, ως προς τις τιμές δηλαδή μπορούν να προτείνουν οι εταιρείε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν μέσα στην Ευρωζώνη αλλά και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ζήτημα όμως και των ε, ταξιδιών για επιχειρηματίες. Δηλαδή κινδυνεύουν και οι επιχειρήσεις να πληγούν όπως ακριβώς ο καταναλωτής, ο ιδιώτης καταναλωτής όταν υπάρξουν ε, ε, προβλήματα στις αερομεταφορές. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Για να είναι η Ευρώπη η γη της υπεροχής και της ακρίβειας της αερομεταφορές και της ε, ικανοποιητικής αποζημίωσης και της εξέβρεσης των κατάλληλων και εναλλακτικών λύσεων. Γιατί θα ήταν πολύ καλό, επί παραδείγματι, να ε, προσφέρεται η εναλλακτική λύση, που ενδεχομένως να μην είναι καν αεροπορική, αλλά μια άλλη μορφή μεταφορών. Για να γίνει λοιπόν η πρώτη στην, ε, εξυπηρέτηση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών η Ευρώπη, θα πρέπει να προσφέρουμε και για τις επιχειρήσεις αυτήν την ε, την προστασία. Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται μέσα αυτή τη ε, λειτουργία της εσωτερική αγοράς να αποστέλουν τους συνεργάτε, το προσωπικό τους, δεξιά-αριστερά ανά την Ευρώπη και βέβαια χρειάζονται την ίδια προστασία. Κύριε Μάιερ, είμαι πεπισμένο ότι θα συνεχίσουμε με τις προτάσεις σα την επικοδομητική συνεργασία και πάλι ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Βιλάνιν Αλλά παρακαλώ με συντομία γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Ευχαριστώ και Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του γνωμοδότηση. Συμφωνώ, δεν πρέπει μόνο τις λεπτομέρειες να προσέξουμε, αλλά και να διευκολύνουμε, να απλοποιήσουμε το κείμενο γενικότερα, για να μην αναφέρει συνέχεια άλλους κανονισμούς και οδηγίες. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε, στις βασικές μας, μας ιδέες. Εγώ προσωπικά βρίσκω ότι το θέμα έχει μένει συζητηθεί πάρα πολλές φορές αλλά δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Οι επιβάτες ακόμη δεν πληροφορούνται σωστά για τα δικαιώματα που έχουν και οι αεροπορικές εταιρείες κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας των θέσεις. Και αυτό δεν το λέω γιατί είμαι κατά των αεροπορικών εταιριών καθεαυτών, όχι βέβαια. Και αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα. Λέω όμως ότι πρέπει να εξισορροπηθούν οι δύο πλευρές. Πρόκειται για τις δύο πλευρές ενός συμβολέου αν υπάρχουν δικαιώματα που δεν εφαρμόζονται ή δεν τα γνωρίζει ο επιβάτης, τότε πρέπει να υποβάλλονται κυρώσεις. Ε, δεν έχω ακόμη κατασταλάξει ως προς τις τρεις ή πέντε ώρες. Πρέπει να μιλήσω με τα μέλη της ομάδας μου πρώτα. Αλλά αυτά που προτείνει ο κύριος Μάγερ νομίζω κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Όσο για τις αλλαγές στο παράρτημα 1 για τις εξαιρετικές συνθήκες, δεν πρέπει να αλλάξουμε νομίζω τη σειρά που έχει ο κατάλογος. Τώρα, οι αλλαγές για το παράρτημα 2. Μιλάμε για ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα. Συμφωνώ με τον κύριο Μάγερ ότι η αναφορά στο ευρώ είναι σωστή. Τώρα, για το σημείο 9, άρθρο 9. Εκεί μιλάμε για το κόστος διανυκτέρευσης και η Κομισιόν προβλέπει 100 ευρώ. Αναρωτιέμαι, ποιος το αποφάσισε αυτό, τον αριθμό τα 100 ευρώ. Γιατί το αν θα είναι 100 ή 150 εξαρτάται από τον προορισμό. Ε, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν την Κομισιόν ποιος αποφάσισε το ποσό αυτό κατά αποκοπή των 100 και για το 4 εισιτήρια επιστροφής εάν ένας επιβάτης έχει πληρώσει για εισιτήριο μετεπιστροφής γιατί τότε πρέπει πρώτα να εκτελέσει την πτήση ΑΛΕ πριν να μπορεί να χρησιμοποιήσει την πτήση ρετούρ. Δεν πρέπει να έχει σημασία η σειρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ριά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο όπω ζητήσατε. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, πρέπει το τελικό αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά σαφές και νομίζω ότι είναι σημαντική η συμβολή του κυρίου Μάγερ με την έκθεσή του γιατί ξέρω ότι υπάρχει ε, στιγνός ανταγωνισμός ε, στις ευρωπαϊκές ε, γραμμές και έτσι αυτό δημιουργεί σε ασάφεια στις διαδικασίες και θέλει να αποφύγει ο κλάδος και το ενδεχόμενο τέτοιων καθυστερήσεων ε, σε διαπραγματεύσει και διακανονισμού με του επιβάτε. Όταν όμω υπάρχουν τέτοιε ασάφειε και βεβαιότητε, αυτό θα γίνει. Και τότε οι αεροπορικές γραμμές θα πάνε πολύ μακριά για να καταφέρουν να μην πετύχουν και να μην, να μην πληρώσουν, συγγνώμη, να μην καταβάλουν αποζημιώσεις. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά και τον κατάλογο να είναι ω δυνατόν πιο ξεκάθαρος. Ε, ο κατάλογο των εξωτερικών αυτών συνθήκων είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε ανοίγματα για ε, εξαιρέσει και για ασαφείς έννοιες. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Δεύτερον, η μέρημνα θα είναι πιο, πιο σημαντική από ότι η αποζημίωση. Γιατί όταν υπάρχει πραγματικό κόστος ε, ή ζημία, τότε πράγματι πρέπει να λάβει κάποιο αποζημίωση. Όμως ε, ε, υπάρχει και αυτή η συζήτηση με τα καταπο, ποσά. Έχουν δημιουργηθεί και κάποιες ε, ε οργανώσεις, οι λεγόμενες ε, claim organizations που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα ακριβώ, με την αποζημίωση κάποιων τέτοιων ισχυρισμών και με ευθύνη και των αεροπορικών ε, αερογραμμών γιατί δυσκολεύουν αυτή τη διαδικασία υποβολής παραπώνων όμως ε, είμαι αρκετά ευέλικτο ό,τι αφορά τα δικαιώματα αποζημίωση, Όχι όμω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ε, για τη μέρημνα. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, καθυστέρηση, ακύρωση... Είναι σημαντικό να μην συμβεί αυτό που έγινε σε μένα στο Μαϊάμι, όπου ξαφνικά βρέθηκα σε ένα τεράστιο χάο, κανένα δεν ξέρει τι συμβαίνει, κανένα δεν ξέρει ε, αν δικαιούμαστε διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο ή όχι, σε ποιο ξενοδοχείο. Πραγματικό και απόλυτο χάος. Και Στη συνέχεια η αεροπορική γραμμή το διόρθωσε. Όμως αυτές τις δύο ημέρες πραγματικά ε, μας κατέστρεψε τις διακοπές, γιατί ήταν και στο τέλος των διακοπών. Η μέρη λοιπόν θα, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά καλά στοιχεία εδώ και εγώ έχω κάποιες τροπολογίες για, για τη διάρκεια και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που θα πρέπει να παρέχει η αεροπορική. Συμφωνώ και με αυτό που υπόθηκε για το ποσό των 100-150 ευρώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξαρτηθεί από τον τόπο, γιατί οι τιμέ διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Όμως ξέρω πολλούς αερολιμένες όπου κανείς δεν μπορεί να βρει δωμάτιο για 100 ευρώ σε καμία περίπτωση. Τα 150 είναι σίγουρα ένα πιο ρεαλιστικό ποσό. Σίγουρα θέλουμε από την ομάδα μου να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά καλή η βάση και θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε κάτι παρετέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στήλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μάιερ και τον κύριο Μπαχ. Νομίζω ότι αυτή η συνεργασία σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντική να γίνει σωστά πρέπει. Ο κύριος Βοσφόγ νομίζω ανέφερε ότι και εμείς έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα θετικών και αρνητικών εμπειριών με την εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος. Υπάρχουν καλές προθέσεις στο νομοθέτημα, όμως η εφαρμογή του σε πολλές περιπτώσεις ε, υπολείπεται. Κάποιες φορές ε, έχω ακούσει για περιστατικά όπου καθυστέρησε πτήση για 10 ώρες χωρίς να ε, λάβει αποζημίωση. Γιατί εδώ όταν ε, κλείνει κάποιο συστήριο μέσω ενός πακέτου, οι υπεύθυνοι που είχαν αναλάβει αυτό το πακέτο άλλαξαν την εταιρεία ε, που θα τον πήγαινε στον προορισμό του. Και μετά υπάρχει αυτή η αμφισημία. Ποιο έχει την ευθύνη, αυτό που έκλεισε το εστήριο ή η αεροπορική ε, γραμμή που μετά είχε τα προβλήματα. Τα προβλήματα. Πολλοί ψηφοφόροι μας γράφουν για τέτοια περιστατικά με αρνητικές εμπειρίες και είναι καλό που μας, ε, τις μοιράζονται αυτές τις εμπειρίες μαζί μας και μας ενημερώνουν για να φροντίσουμε να μην ξανασυμβούν τέτοιου ε, περιστατικά. Αυτό που ανέφερε συνάδελφος προηγουμένως για την ευθύνη, ε, την υπευθυνότητα σε τέτοιες ε, περιπτώσεις είναι σημαντικό. Εγώ είχα μια θετική εμπειρία. Μια φορά που πήγαινα στο Τρασβούργο, ε, ξέρετε τι συμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις, απευθείας μας δώσανε τα κουπόνια για την ε, για διατροφή και το, και το καθεξής αλλά ξέρουμε ότι αρκετές αεροπορικές εταιρείες τα πάνε πολύ καλά. Δεν είναι όλα αρνητικά. Γιατί λοιπόν κάποιες αεροπορικές συμμορφούνται με το πνεύμα του νόμου και άλλες ε, το αποφεύγουν. Εφόσον τα συζητούμε όλα αυτά, είναι σημαντικό να γίνεται ανταλλαγή των πρακτικών και να προσθέτουμε και τις δικές μας ε, θετικές εμπειρίες και όχι να έχουμε τέτοια περιστατικά όπως αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ για τους δύο για τη συνεργασία και ελπίζω να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα για να δείξουμε και στους ψηφοφόρους μας ότι όταν ξέρουμε παιδεία όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν πρωτοείδα της τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπα χρειάζεται περισσότερο δίκαιο, περισσότερα δικαιώματα, περισσότερη προστασία του καταναλωτή στην υπόθεση αυτή. Βλέπω όμως με χαρά ότι ο εισηγητής, οι δύο εισηγητές έχουν ε, την πρόθεση να εισαγάγουν πολλές τροπολογίες προς τη σωστή κατεύθυνση. Βλέπουν ότι είναι περίπλοκη η πρόταση της Επιτροπής. Ε, όροι όπως μέγεθος του αεροπλάνου, στους οποίους δεν έχει καμία ε, επίδραση ο ε, επιβάτης ή το αν έχει 90 ή 91 επιβάτες είναι πράγματα πρέπει να φύγουν και γι' αυτό χαίρομαι για τις προτάσεις σας. Στην αναλογικότητα της αποζημίωσης έχω μια ερώτηση, μια πρόταση που ε, υποστηρίζει ο κύριος Μάιερ και ο κύριος Μπαχ μας λέει ότι είναι μάλλον υπερβολικά περίπλοκη. Τότε γιατί ε, ε, θα έχουμε την εικόνα να, έχω, να λαμβάνουν διαφορετική αποζημίωση επιβάτες με την ίδια καθυστέρηση. Δεν θα σημαίνει αυτό μια στάση, όχι ουδέτερη απέναντι στον επιβάτη, μια στάση που θα εξαρτάται από το μέγεθος του πορτοφολιού του. Αλλά από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι λαμβάνουμε υπόψη ε, ζημία, οικονομική ζημία, η οποία δεν εξαρτάται όμως από το τίμημα του εισιτηρίου. Και γι' αυτό, κύριε Μάιερ, θα σας παρακαλούσα να εγκαταλείψετε αυτή την ιδέα της αναλογικότητας, η οποία μου φαίνεται και υπερβολικά ε, γραφειοκρατική και Εξάλλου μπορεί να οδηγήσει του επιβάτε σε μία πλάνη. Δεν θα μπορούν τα Έλληνα να γνωρίζουν τι είδου δικαιώματα έχουν. Μπορεί να μην ξέρουν με βάση ποια ταρήφα, με βάση ποια τιμολογιακή κατηγορία έχουν πληρώσει το ειστήριό του και τι μπορούν να διεκδικήσουν. Είναι πολύ περίπλοκο. Ευχαριστώ. Έχουμε τον κύριο Κόλσον της Επιτροπής. Θα παρακαλέσω αν έχει την καλοσύνη να μας κάνει σχόλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την έκθεση. Περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες διευκρινήσεις επί πολλών ζητημάτων και το χαιρετίζουμε. Συμφωνούμε με κάποιες από τις προτάσεις όπως αφορούν τις καθυστερήσεις ε, ε, στην επίσταση στο αεροδιάδρομο. Νομίζουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν ήταν αρκετά καλή από αυτή την ε, πλευρά και θα ήταν καλό να το εξετάσουμε. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω τέσσερα σημεία επιφύλαξη που έχει η Επιτροπή σε σχέση με την έκθεση και θα μείνω στα ζητήματα που αφορούν αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Για να μην περάσουμε στα ζητήματα που αφορούν την έκθεση του κ. Μπακ. Πρώτον, τροπολογία 29. Με αυτή την ε, τροπολογία ο εισηγητής προτείνει να αρθεί η καθυστέρηση των δύο ε, ωρών για την ε, παροχή μέρημνας σε περίπτωση καθυστέρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες δικαιούνται με μετά από καθυστέρηση ακόμα και ενός λεπτού. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι υπερβολικό. Δεύτερο, τροπολογία 42. Εκεί προτείνεται να περιοριστεί η αποζημίωση στην ε, αξία ε, του εισιτηρίου. Η επιλογή της Επιτροπής ήταν να μην ε, τροποποιήσει το ποσό της αποζημίωσης, αλλά να αυξήσει το όριο της ε, καθυστέρησης από τις 2 στις 5 ώρες. Έτσι η πρόταση διαφέρει από την έκθεση. Όπως και να έχει, θα πρέπει να αποφύγουμε ε, αυτή την πρόταση σε σχέση με την άρνηση επιβίβασης. Γιατί αν υπάρχει αποζημίωση ανάλογική, ανάλογη ε, της τιμής του εισιτηρίου σε ό,τι αφορά την άρνηση επιβίβασης, τότε η αεροπορική θα ενδεχομένως να αρνηθεί ε, επιβίβαση στους επιβάτες που έχουν αγοράσει φθηνότερο εισιτήριο, αν θέλετε. Δεν νομίζουμε λοιπόν ότι η αποζημίωση βάσει της τιμής ή επί ποσοστού της τιμής ότι είναι μια κατάλληλη και ακριβής ε, μέθοδος σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης. Τρίτο, ε, για την τροπολογία 53. Εδώ η συγητής ε, διαγράφει την απαλλαγή από τη διαμονή για τις περιφερειακές πτήσεις ή τοπικές πτήσεις. Αυτή η εξαίρεση που βρισκόταν στην πρόταση της Επιτροπής είναι σημαντική γιατί Εάν δεν υπάρχει αυτή η εξαίρεση στον κανονισμό, αυτό σημαίνει δυσανάλογο βάρος για τις ε, μικρές ε, περιφερειακές ε, εταιρείες που αφορούν πτήσεις κάτω των 250 χιλιόμετρων και με ε, λιγότερες από 80 θέσεις. Τέταρτο, Τροπολογία 66. Εδώ η συγκητής ε, προτείνει το ADR, ε, ο μηχανισμός ε, διακανονισμού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες για να δοθεί απάντηση. Αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 8α της οδηγίας ADR του διακανονισμού, η οποία υιοθετήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες. 2013 κάθετος 11 που δηλώνει ρητός ότι ο διακανονισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή σε περίπτωση ιδιαίτερα περίπλοκων υποθέσεων. Επομένω, δεν είναι δυνατόν ε, βάσει τη οδηγία να περιοριστούμε στι 90 ημέρε. Αυτό αντιβαίνει στην οδηγία 2013 11, η οποία δηλώνει ξεκάθαρα στο άρθρο 3 ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί άλλη νομοθεσία, άλλο νομοθέτημα να ε, να υπερισχύσει ε, αυτής. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ε, να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 9η Οκτωβρίου στις 12 το Να δώσουμε και πάλι το λόγο στον εισηγητή για δύο λεπτά να δώσει κάποιες πρώτες απαντήσεις και θα έχουμε πολύ καιρό στη συνέχεια. Ευχαριστώ και αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και την υποστήριξη. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Σημαντικό για μένα είναι βέβαια να είναι σαφή η κατάσταση ω προ τα χρονικά όρια, τι προθεσμίε, ε, τι αποσκευέ ή χειραποσκευέ, όλα αυτά τα οποία μπορούμε να ε, ορίσουμε για να αποφεύγουμε την, ε, καταφυγή, την προσφύγη στα δικαστήρια. Οι αεροπορικές εταιρείες, αγαπητοί συνέλφοι, υπολογίζουν το χρόνο των πτήσεων τους, μάλλον τις πτήσεις που μπορούν να προσφέρουν, κατά τρόπο ώστε, εάν πωλήσουν και το αλέ και το ρετούρ, να μην έχουν απώλειες. Πολύ καλά. Σωστό είναι αυτό. Εάν λοιπόν κάποιος πάρει και το αλέ και το ρετούρ, δεν έχει απώλειες οι αεροπορικές εταιρείες και ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσουμε εμείς την πτήση του πήγαινε, δεν έχει χάσει τίποτα η αεροπορική εταιρεία γιατί τον έχουμε πληρώσει, το ειστήριο το έχουμε πληρώσει δεν έχει λόγο μετά να μας αρνηθεί την επιστροφή. Δεν ζητάω να μου κρατήσει τη θέση μου, μπορεί να ξαναπουλήσει την ίδια θέση άλλων επιβάτη. Δεν μπορεί όμως να κερδίσει και παραπάνω αρνούμενη την ε, επιβίβασή μου στην ε, πτήση της επιστροφής. Νομίζω και αυτό μπορούμε να το περιορίσουμε ή πρέπει να το περιορίσουμε. Υποχρέωση και ενημέρωση. Πολύ σωστό είναι αυτό, είναι πολύ σημαντικό είναι απαραίτητο να προσφέρεται και στις 24 γλώσσες, γιατί προφανώς εάν έχω φτάσει σε μια χώρα της οποίας δεν γνωρίζω την γλώσσα, τι να κάνω όσα ε, δελτία πληροφόρηση να μου δώσουν αν δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα. Άρα πρέπει να είναι διαθέσιμη και στις 24 γλώσσες. Ο ε, περιορισμός της αποζημίωσης στην τιμή του εισιτηρίου. Να σας πω, εγώ όμως λέω το εξής στο σύνολο της τιμής του εισιτηρίου μαζί με την επιπλέον επιβάρυνση για αποσκευές κτλ. Ξέ, και αυτό ξέρετε δεν είναι ιδιαίτερη επιβάρυνση γραφειοκρατική για τον επιβάτη, ξέρει τι έχει πληρώσει. Πλήρωσε 100 ευρώ, πλήρωσε 25 ευρώ, ό,τι είναι ξέρει τι έχει πληρώσει. Είναι πολύ ορατό πάνω στο, στο τιμολόγιο και την απόδειξη που έχει πάρει. χρονοθυρίδες και δύο ή πέντε ώρες ε, στον ε, διάδρομο απογείωσης. Ε, κοιτάξτε να σας πω, όταν έχουμε χιονοθύελες και όταν πρέπει να γίνει η ειδική διαδικασία για το ξεπάγωμα των αεροπλάνων ή να περιμένουν να περάσει μία μπόρα, δεν μπορεί να εξαρτηθεί η η πτήση από την απέτηση για τις δύο ή τις 5 ώρες, είναι λογικό ότι ο πιλότος θα περιμένει να είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες. Οι δύο ώρες νομίζω ότι αρκούν. Και εν τέλει, στις προτάσεις της Επιτροπής για την άμεση παροχή εξυπηρέτησης. Είπε πολύ σωστά η συναδελφός ότι όταν βλέπει ότι μπορεί να έχει μία καθυστέρηση μία-δύο ωρών ε, στο Στρασβούργο, τη δώσαν ένα σαντουιτσάκι κτλ. Ναι, βεβαίω. Δεν μπορώ να περιμένω να περάσουν δύο ώρε για να μου δώσουν ένα ποτήρι νερό να πιω. Ούτε και πρόκειται αυτό να οδηγήσει σε πτώχευση τη ε, εταιρεία. Κάποια θέματα λοιπόν, ακόμα όπως βλέπω, πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε, αλλά μπορούμε να καταλήξουμε σε πολύ καλές και λογικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστούμε. Τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική περίθαλψη. Θα πάρουμε τις τροπολογίες για τα δικαιώματα των επιβατών. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ερικόγιαν Περές, αλλά δεν τη βλέπω εδώ. Μήπως υπάρχει κάποιος που την αντικαθιστά. Ναι. Ο κύριος Γκάστης Ραμών. Εντάξει, έχετε το λόγο. Λοιπόν. Το Αντικαθιστώ τη συνάδελφό μου κυρία Εργογέν που κολλείεται σήμερα να παραστεί για προσωπικούς λόγους. Και μου ζήτησε να σας πω τις απόψεις της για την έκθεση αυτή της ηλεκτρονικής περίθαλψης 2012. Πρώτον, ευχαριστεί τα μέλη που κατέθεσαν τροπολογίες και ιδιαίτερα τους Σκιώδης για τη συνεργασία τους. Επίσης έχει λάβει 28 τροπολογίες που τονίζουν μερικά θέματα πιο πολύ όπως την προώθηση του ρόλου του υγειονομικού προσωπικού και οργανώσεων καθώς και των ιδίων των ασθενών για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού ηλεκτρονικής περίθαλψης ή ήτα περίθαλψης όπως λέμε. Η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ χωρών μελών τονίζεται επίσης η ανάγκη Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση ηλεκτρονικών υπαλλαγιστών μπορεί επίσης να συμβάλλει. Έχει καταθέσει έξι συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουν διανεμηθεί στις πολιτικές ομάδες και που καλύπτουν όλες τις άλλες. Νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε πλήρη υποστήριξη στην τελική ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Πιέτη Κάινεν που είναι σκιώδης του ΕΛΚ. Ευχαριστώ καταρχήν, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία Γίνονται εδώ μεγάλες πρόοδοι για το θέμα αυτό της ήττα υγείας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την υγεία ιδιαίτερα, αλλά και τις καινούργιες βιομηχανικές δυνατότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Εμείς στο ΕΛΚ Αναμένουμε ανυπομόνως το, τη μελλοντική πράσινη βίβλο για το θέμα αυτό και καταλαβαίνουμε ότι η Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για θέματα προστασίας δεδομένων, πρόσβασης στα δεδομένα, πληροφόρησης υγειονομικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα τη δυνατότητα δημιουργίας πανενοσιακών κέντρων χορήγησης τέτοιων υπηρεσιών. Γενικά το ΕΛΚ είναι σχετικά ικανοποιημένο με τις συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά υπάρχουν ακόμη δύο θέματα που θέλουμε να θίξουμε και ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, η συμβιβαστική τρία που μιλάει για την ανάγκη μετεκπαίδευσης των ανθρώπων στα ηλεκτρονικά. Η αρχική μας τροπολογία 10 βασιζόταν στην προσβασιμότητα. Τα σύστηματα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους. Όταν σχεδιάζουμε λοιπόν ένα σύστημα πρέπει να το λαμβάνει ήδη υπόψη του από την αρχή αυτό. Να σκέφτεται τους λιγότερο μεμορφωμένους, τους αναπήρους και να είναι εύκολη η πρόσληψη του χρήστη. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Μιλήσαμε για την προσβασιμότητα γενικότερα των ιστοσελίδων, αλλά είναι και αυτό θέμα ισότητας. Ελπίζουμε λοιπόν η τροπολογία μας 10 να ληφθεί υπόψη στις συμβιβαστικές. Ένα άλλο θέμα είναι η συμβιβαστική έξι. Στο ΕΛΚ εμείς δεν θεωρούμε ότι η αιτήσια αναφορά προσθέτει τίποτε σημαντικό. Τονίζουμε περισσότερο την ανάπτυξη του ίδιου του προγράμματος και ζητούμε αναφορά κάθε δύο χρόνια Αυτά ήθελα να σας πω. Τα υπόλοιπα καλύπτονται σωστά. Τα προσωπικά αρχεία υγείας πρέπει να υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή και να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι χρήστες. Με μεγάλη προστασία βέβαια για να μπορεί να έχει πρόσβαση μόνον ο ενδιαφερόμενος. Να έχουμε δηλαδή μια ευρύτερη αντίληψη του θέματος από την αρχή ήδη του σχεδιασμού του συστήματος. Και ο ρόλος της Κομισιόν να είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και η διασφάλιση της συνδυαστικότητας των διαφόρων συστημάτων. Για την προστασία των δεδομένων είναι γνωστό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Παρβάνοβα από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την εισηγήτρια και όλους τους άλλους συναδέλφους. Θέλω απλώς να αναφέρω τα κύρια θέματα όπου δεν έχουμε ακόμη πετύχει συμβιβασμό. Ευτυχώς το σύνολο των τροπολογιών είναι μόνο 28, δεν ήταν λοιπόν πάρα πολλές, υπάρχουν 6 συμβιβαστικές. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων υποστηρίζουμε και τις 6, ιδιαίτερα το ότι πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες ως προς το τι πρέπει να βελτιωθεί. όπως η μείωση των ανισοτήτων κλπ. ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης. Επίσης, εκείνες που αναφέρουν στην δημιουργία τραπεζών δεδομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αποθήκευση των προσωπικών υγειονομικών δεδομένων των χρηστών. καθώς και τη φροντίδα να μην υπάρξει άνηση μεταχείριση και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη διαμεθοριακή συνεργασία και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο. Η τροπολογία 7 της κυρίας Πέρες θα έλεγα ότι το θέμα της αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί περισσότερο στην Επιτροπή αν συμφωνήσουμε από εδώ θα περάσουν πιο εύκολα οι τροπολογίες μας και στην κύρια επιτροπή που είναι η περίφ. Ευχαριστώ. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι το λόγο. Σκιώδης. Γι' αυτό θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρεμπέλος από την Κομισιόν να σχολιάσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια. Σημείωσα μερικά πράγματα. για την πράσινη βίβλο προβλέπεται να εγκριθεί πριν το τέλος του χρόνου και να γίνει και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για να έχουμε ακούσει όλες τις απόψεις Είναι προγραμματισμένο λοιπόν αυτό. Τι άλλο είχα πει για το e-porting. Προσπαθήσαμε, reporting μάλλον, προσπαθήσαμε να τα σταθμίσουμε και αυτά και θέλουμε η, η να μπορέσει να ακολουθεί κάπως τα υπόλοιπα μέτρα που λαμβάνουμε και για την επιμόρφωση για να μην υπάρχουν άνισες άνοιχη μεταχείριση και να γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και αυτό μέσω του δικτύου ή τα Υγείας θα γίνει ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να κάνουν ακόμη περισσότερες ανταλλαγές εμπειριών Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκαρσές Ραμών για να καταλήξει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι πολύ ικανοποιημένο που βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση μεταξύ των πολιτικών αμάδων. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι για τις συμβιβαστικές 3 και 6. Το πρωί, λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίασή μας, έγινε μια νέα διατύπωσή τους που με προσπάθεια συμπερίληψης και των αντιδράσεων του ΕΛΚ και με αυτή την αλλαγή νομίζω ότι θα μπορέσει και το ΕΛΚ να τις δεχτεί επίσης προς την Κομισιόν θα ήθελα να είπω ότι είναι καλά τα νέα ότι η πράσινη βίβλος θα δημοσιευτεί πριν τα τέλη του έτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει την Δευτέρα. Επόμενο θέμα λοιπόν πρόσβαση αγαθών τρίτων χωρών στην ενωσιακή αγορά δημοσίων προμηθειών. Φρανκ Έγγεν είναι ο εδώ είναι και αυτός και έχει και το λόγο. Στην On the, uh, market access... Uh, Στα αγγλικά καλύτερα. Έχουμε διάφορα θέματα αρχής. που δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε. Θα σας πω λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Θα σας πω ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τα δικά μας θέματα από την ώρα που έγινε η σύνταξη και αναλάβαμε τα θέματα των οποίων επιλαμβανόμαστε και θεωρώ ότι είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Μου φαίνεται παράξενο να συζητούμε ή να διαπραγματευόμαστε ζητήματα ε, που έρχονται με τροπολογίες και που ξεπερνούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Επίσης, με κάποιοι συνάδελφοι μεταξύ των οποίων και οι εξαριστερών μου, προσπαθούν να απορρίψουν όλη την πρόταση. Πολύ καλά. Έχουν κάθε δικαίωμα, αλλά δεν συμφωνώ. Και ως εκ τούτου απορρίπτω η αδίποτε τέτοια πρόταση. Δεν αφαιρώ το love ή το like από τους ε, φίλους που ενδεχομένως ακολουθήσουν τη στάση αυτή, αλλά δεν ακολουθώ αυτές τις προτάσεις. Ε, επί της ουσίας, στο θέμα αυτό, όπως ε, ξέρετε, έχουμε διαφορές απόψεων μεταξύ Γάλλων και Γερμανών. Και εγώ τίνω να ακολουθώ μάλλον τους Γάλλους, χωρίς να σημαίνει ότι προσυπογράφω οτιδήποτε μου προτείνουν, αλλά τουλάχιστον για την ουσιαστική αμοιβαιότητα και τα συναφή, θα συμφωνούσα και νομίζω ότι μπορούν να προσφέρουν προσθέμενη αξία στο κείμενό μας. Ραφαέλε, Ραφαέλε, μα όλη αυτή η αντιγραφή και επικόλυση των ε, αφύσικα χαμηλών προσφορών, ε, προφανώς και για λόγους, αφού έχει ήδη απορριφθεί σε προηγούμενη πρόταση, για λόγους και συνοχής, δεν πρόκειται να υποστηριχθεί. Όλες λοιπόν οι προτάσεις που στόχο έχουν να φέρουν σε συνέπεια την ε, πρόταση αυτή με την πρόταση για τις δημόσιες προμήθειες και τις αναθέσεις που βεβαίως απαιτείται Αυτά λίγο πολύ είχα να πω. Περιμένω να ακούσω τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι. Καλώς ευχαριστώ. Σκιώδης ηγητές, η κυρία Βάιλερ, πρώτη εκ Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Κύριε Έγκελ, αγαπητοί συνάδελφοι, Όποιος έχει ρίξει μια ματιά στις ε, τροπολογίες θα έχει διαπιστώσει ότι και οι σοσιαλδημοκράτες ε, βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Και σα το λέω απερίφραστα, είναι γνωστό άλλωστε, ότι στην ομάδα μας άλλοι τίνουν προς τις θέσεις της Γαλλίας και της Νότιας Ευρώπης, άλλοι προς τη Βόρεια Ευρώπη, υποστηρίζουμε γενικά τις, υποστηρίζουν γενικά την πρόταση, άλλοι και άλλοι όπως εγώ και κάποια άλλοι είναι πιο επιφυλακτική Και είμαι πιο επιφυλακτική για το εξή: ότι βλέπω ότι περιορίζεται χωρίς η αιτιολόγηση η λειτουργία της αγοράς. Με τη ρύθμιση παραδείγματι των ε, ε, ηλιακών ε, κύψελών των φωτοβολταϊκών συστημάτων ε, που προέρχονταν από την Κίνα, το είδαμε αυτό ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Και εδώ, κύριε Έγγελ, νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ορισμένα ζητήματα, εφόσον πρόκειται απλώς για γνωμοδότηση, να τα κρίνει μόνο η Ολομέλεια. Και γι' αυτό θα περιοριστώ τώρα μόνο σε αυτά τα οποία πραγματικά μας ενδιαφέρουν, κανόνες που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές συνθήκες και ε, προδιαγραφές ε, εργασίας και με τις συνθήκες εργασίας. Αυτά λοιπόν, τα οποία ήδη έχουν εκριθεί σαν νομοθετήματα για λόγους συνέπειας θα πρέπει να τηρηθούν και εδώ και ιδιαίτερα σε σχέση με το διεθνές εμπόριο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ομάδα μου. Δεν μπορούμε να λησμονήσουμε στους τομείς αυτούς τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία της απασχόλησης των εργασιακών σχέσεων. Και από την άλλη, μεγάλο ερωτηματικό διατυπώνω για το κατά πόσο χρειάζεται το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλε. Με ξεχάσατε, Πρόεδρε, πριν δεν με είδατε, αλλά δεν ε, αντέδρασα γιατί δεν είναι τόσο σημαντικά τα θέματα. Τώρα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογία για απόρριψη και θα ψηφίσουμε αποφασιστικά για να απορριφθεί αυτή η πρόταση και πιστεύω ότι όλοι μας εδώ, οι εκπρόσωποι της ομάδας μου στην Επιτροπή αυτή συμφωνούμε. Δεν είναι επαρκής για να δώσει βάση και αιτιολόγηση για μια τέτοια οδηγία η πρόταση Επιτροπή. Είναι σφαλμένη η επιλογή και η κατεύθυνση αυτής της οδηγίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε διεθνές εμπόριο και όχι με δημόσιες συμβάσεις. Εάν λοιπόν φορτώσουμε τις δημόσιες συμβάσεις ε, στο θέμα αυτό, τότε δημιουργούμε τέτοιες πιέσεις οποιονδήποτε εργολάβο θέλει να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συμβάσεις που, δεν θα, που θα εξυπηρετήσουμε τον ακριβώς αντίθετο σκοπό από αυτόν που δεν θα εξυπηρετούμε. Ευχαριστώ. Καταψηφίζουμε λοιπόν αποφασιστικά. Καλώς, ευχαριστώ. Κύριε Μακλάρκιν, ECR. Ευχαριστώ, αγαπητή Σάλφη, κύριε Έγκελ. Όπως ξέρετε, εγώ αντιτίθεμαι στην πρόταση αυτή, στο σύνολό τη. Βλέπω ότι και άλλοι συνάδελφοι ίσως να δυσκολεύονται να την ε, υποστηρίξουν στο σύνολό τη. Νομίζω ότι μη τι άλλο δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλες τροπολογίες για απόρριψη αιτιολογείται και η δική μας η επιφυλακτικότητα ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ την κυρία Ρούλε και την συγχαίρω για την αποφασιστική της καταδίκη της προτάσεως στο συνολό και την μπορεί, <laughs> έχοντας καταλήξει στο ίδιο, στο ίδιο αποτέλεσμα, να ερχόμαστε από διαφορετικές ε, αιτιάσεις. Το κύριο θέμα λοιπόν, το άρθρο 6 που δίνει τη δυνατότητα αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις ε, προμηθευτών από τρίτες ή οικονομικών φορέων από τρίτες χώρε. νομίζω θα αποβείς ε, βάρος των ε, επιχειρήσεών μας, της ενιαίας αγοράς, θα περιορίσει τον ελεύθερο και θεμητό ανταγωνισμό, θα αυξήσει τις τιμές. Είναι εσφαλμένη η επιλογή αυτή και κυρίως σε περίοδους οικονομικής αστάθειας. Ελπίζω να με υποστηρίξουν, να με κατανοήσουν καταρχάς τα επιχειρήματα αυτά και να με υποστηρίξουν και οι λοιποί συνάδελφοι για να αποσυρθεί, για να διαγραφεί το άρθρο αυτό. Επίσης την πρόταση για ασυνήθιστα ή αφύσικα χαμηλές προσφορές. Όχι, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την ε, διάρκεια της διαδικασίας, όχι να επιβάλλουμε ακόμη περισσότερους όρους αυτές τις διαδικασίες των ε, συμβάσεων, των διαγωνισμών, αλλά να σας το πω γενικά, απλώς δεν μου αρέσει αυτή η πρόταση. και βλέπω ότι και η κατουσίαν αρμόδια επιτροπή έχει η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή έχει μια όλο και εντυνόμενη τάση να απορρίψει την πρόταση συνολικά. Έχουμε λοιπόν αρκετά εργαλεία, έχουμε την τροποποιημένη οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες, έχουμε τις δημόσιες συμβάσεις, έχουμε τις δύο οδηγίες για την εσωτερική αγορά. Ε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβαρυνθεί το νομοθετικό μας πλέγμα και με άλλο ένα νομοθέτημα. Ευχαριστώ. Κύριος Βαλτασάρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από μία πιο εις βάθος ανάλυση. Εδώ που πρέπει να αναλύσουμε τις, ε, τα πεδία αντιπαράθεσης μεταξύ διαφόρων κέντρων και νομίζω ότι αν κάποιος πει ότι υπάρχουν δύο τελικά Ευρώπες, μάλλον θα έχει δίκιο. Γιατί βλέπουμε ότι και στην, ε, στο σήμα καταγωγής ή προέλευσης και στις δημόσιες ε, προμήθειες και στην αμοιβαιότητα για τις δημόσιες συμβάσεις βλέπουμε ότι άλλα λέει μισή Ευρώπη και άλλα η άλλη μισή. Και δεν καταφέρουμε να συγκεράσουμε τις διαφωνίες μας. 12 δισεκατομμύρια, μας λέει η Επιτροπή, χάνονται από αυτή την υπόθεση και κυρίως στους τομείς εκείνους τους οποίους είχαμε στο παρελθόν τις ηγετικέ θέσεις, δηλαδή στην κατασκευαστική και στους σιδηροδρόμους. Έτσι, και αν μπορούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να διαφυλάξουμε θέσεις εργασίας, θα πρέπει να το πράξουμε. Το 2003 οι Κινέζοι εισήγαγαν παραδείγματι δικές τους ρήτρε buy local. Αγοράζεις, αγόραζε ε, τοπικά προϊόντα. Επί παραδείγματι δεν μπορεί κανείς να πωλεί στην Κίνα εάν δεν έχει αποδείξει ότι έχει εργάτες ε, Κινέζους ε, ε, χρησιμοποιήσει, ότι έχει μείνει στη χώρα και έχει κάνει επένδυση για πέντε χρόνια και το καθεξής. Το ίδιο και οι Αμερικανοί με το Reinvestment Act ενισχύουν τα προστατευτικά μέτρα. και ζητούν όλο και περισσότερο και επιβάλλουν υποχρέωση για ε, εγχώριες υπηρεσίες και προϊόντα. Το ίδιο οι Βραζιλιάνοι, το ίδιο οι Ινδοί και τώρα σε μια περίοδο κρίση εμεί ανοίγουμε τι πόρτε και λέμε «Α, όχι, κάντε ό,τι θέλετε, ε, προσπιστείτε ο καθένα τις δικές του επιχειρήσεις, αλλά εμείς η Ευρώπη είμαστε μια ελεύθερη αγορά, περάστε, κάντε ό,τι θέλετε, πουλήστε τα προϊόντα σας, πουλήστε τα υλικά σας, είμαστε στη διάθεσή σας». Μα πού πιστεύετε ότι θα φτάσετε με αυτή τη συμπεριφορά, πού νομίζετε ότι θα καταλήξει η Ευρώπη και πόσο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει στο δρόμο αυτόν ξεπερνώντας και κατακριμνίζοντας τα εθνικά συμφέροντα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, αλλά για κάποια κράτη μπορεί να είναι συμφέρον να συνεχίζει αυτή η πορεία, αλλά δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει αυτή η πορεία με αυτόν τον τρόπο. Και φτάνω στην ουσία. Άρθρο 6. Εδώ έχουν κατατεθεί τροπολογίες για την διαγραφή του άρθρου 6. Φρανκ, εάν το για κανονισμό που έχει ενισχυμένη ισχύ σε σχέση με την οδηγία και ισχύει αμέσως. Εάν λοιπόν μπορεί να επαληθεύσει τις αρχικές προτάσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες ή αρχή και, δεν, και αν αυτές δεν ξεπερνούν κατά 50% την ε, αξία των ε, αγαθών και ε, υπηρεσιών προσφέρονται. Μα αυτό είναι μια προστατευτική διάταξη, δεν είναι το ελάχιστο για να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη αηφόρο, βιώσιμη, αυτή για την οποία αναγωνιζόμαστε. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην επιχείρηση που θα έρθει να δουλέψει να επιβιώσει. Δεν λέμε ότι πρέπει οι επιχειρήσεις μας να έχουν ε, την ε, φοροανάπτυξη, να πληρώνουν τους φόρους τους, να προσλαμβάνουν κόσμο κτλ. Και μετά λέμε ότι όποιος έχει ε, ανοίξει μια επιχείρηση στον υπόλοιπο κόσμο μπορεί να, φέρνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του υπό οποιαδήποτε συνθήκες ή χωρίς συνθήκες ουσιαστικά στην Ευρώπη. Πού είναι η αμοιβαιότητα μεταξύ αγορών με τα μέτρα αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που ζητείτε είναι στην πραγματικότητα οι άλλοι να ανοίξουν, θα έπρεπε μάλλον να ζητείτε να ανοίξουν τις αγορές τους σε εμάς. Στην πραγματικότητα όμως οι άλλοι, οι τρίτες χώρες, κλείνουν τις αγορές τους. Και σε περίοδο κρίσης εμείς τις ανοίγουμε, ακόμη περισσότερο. Και έρχεστε μετά και μου λέτε να καταργήσουμε το άρθρο 6. Ε, ας καταργήσουμε και το 7, ας καταργήσουμε και όλο το κείμενο. Όλα αυτά στο βωμό ενός το θέμα που είναι η ελεύθερη αγορά. Μα δεν είναι αυτό ελεύθερη αγορά. Αυτό είναι αγορά η οποία θέτει την Ευρώπη σε δυσκολία σοβαρή. Για το άρθρο 7 της προτάσεως. Ιδιαίτερα οι αφύσικα χαμηλές προτάσεις. Εδώ έχουμε αρμοδιότητες κοινέ με την Επιτροπή ΙΜΚΟ και απλώς ζητώ με την τροπολογία μου να εξηγηθούν οι τιμές και το κόστος, εάν είναι πολύ χαμηλότερο, χαμηλότερο κατά 20% ή περισσότερο, από τις λοιπές προτάσεις. Πρόκειται για μια πορεία γραφειοκρατική, η οποία καταδικάζει σε έλλειψη ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις. Κάθε φορά αυτό το επιχείρημα μας ε, προβάλλεται ότι όταν δηλαδή ζητάμε μια περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια στις ε, προτάσεις αυτές τις συμβάσεις, ε, μας λέτε πλήττεται η ανταγωνιστικότητα. Μα δεν μπορούμε να του ρωτήσουμε από πού και ως πού θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά αυτή με λιγότερα λεφτά. Δεν γίνεται έτσι πιο διαφανής η αγορά των δημοσίων συμβάσεων και των προμηθειών. Εάν μπορεί να μας εξηγήσει πού θα βρει τα υλικά και με τι εργάτες θα, θα εκτελέσει το έργο. Δεν είναι αυτή η καλύτερη λύση και όχι το να ανοίγουμε τις θύρες και τις πόρτες τους πάντες, στον υπόλοιπο κόσμο. Έστω λοιπόν, μπορεί να είναι μόνο γνωμοδότηση εδώ το θέμα αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε για να μπορέσει να έχει η Ένωση τα στα κατάλληλα μέσα και να επιβάλλει την πλήρη υλοποίηση των αρχών της διαφάνειας, της αμοιβαιότητας και της ισότιμης μεταχείρισης. Ευχαριστούμε. Πριν ε, δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μου πείτε ποιος από σας θα πάρει το λόγο. Δράτω με της για να σας πω ότι εφόσον έχουμε ακόμα χρόνο, να πω κάτι στον Φρανκ. Με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα. Ε, δεν θέλω να αφαιρθώ σε συγκεκριμένε τροπολογίες είναι περισσότερο πολιτισμικό στοιχείο. Πρέπει να βρούμε μία λύση που να διασφαλίζει την ομοιομορφία στην αγορά, γιατί εμείς πιστεύουμε στην αγορά, αλλά το να απορρίπτουμε κάποια όρια και να σκεφτόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων και όχι μόνο τις υπηρεσίες που παρέχει μία εταιρεία, μπορεί να υπάρξει έλλειψη σαφήνειας και βεβαιότητας σε ό,τι αφορά την αμεβαιότητα μεταξύ κρατών μελών και ομάδων χωρών, αν σκεφτούμε και τις αναδυόμενες οικονομίες. Όλα αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια αγορά καρικατούρα, γιατί δεν έχουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Και άθελά μας μπορεί να καταλήξουμε στα χέρια, θυσία στα χέρια των όσων ε, υποτίθεται ότι στηρίζουν την αγορά, αλλά δεν το κάνουν με το σωστό τρόπο. Θα έχουμε λοιπόν μια αγορά καρικατούρα, όχι μια αληθινή αγορά. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Εγώ πιστεύω πραγματικά στην αμοιβαιότητα. Η μία πλευρά κάνει κάποιες επιλογές, Άλλος ε, κλάδος ε, μπορεί να πρέπει να θυσιάσει κάτι υπέρ της άλλης πλευράς, όμως πρέπει να υπάρχουν ομοιόμορφοι όροι. Αυτό αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και του, και του υπόλοιπου ε, κόσμου, αλλά και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το ίδιο. Τους τελευταίους μήνες το έχουμε εξετάσει, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα χρήζει μια συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει μόνο εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Η κυρία Βάλερ έχει δει το λόγο και μετά η κυρία Γουλερ. Παρακαλώ. Μια σύντομη παρατήρηση μετά από τον πύρινο αυτό λόγο και τη συμβολή του κυρίου Παλτασάρα να υποστηρίξουμε την οδηγία και μια και μιλάμε για πραγματικότητες οικονομικές ε, και οικονομική κατάσταση, εάν η κατάσταση είναι όπως την περιγράφετε εσείς στην Ευρώπη, εάν όντως συμβαίνουν αυτά που λέτε, η Γερμανία δεν θα είχε καμία δυνατότητα να ε, κατασκευάζει μηχανήματα, αυτοκίνητα, χημικά προϊόντα και να πωλεί σε τρίτες χώρες του τρίτου κόσμου, των τρίτων κρατών, της Κίνας και ούτω καθεξής το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτή την τέτοια αυτή, αυτό το, τα προβλήματα ε, εμείς στην Γερμανία καταρχάς αλλά και τα λοιπά κράτη με βιομηχανία της Ευρώπης οφείλεται στο ότι δεν είναι τόσο κλειστές οι αγορές γιατί διαφορετικά αν ίσχυαν αυτά που μας λέτε η Γερμανία θα έχει αρνητική ανάπτυξη. Κυρία Ρούιλε, θα συμφωνήσω και εγώ με την κυρία Βάιλερ Πρέπει τις προτάσεις Επιτροπής να τις κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για τα στοιχεία που προσφέρονται είναι διαφορετικά ακόμα και για το είδος της διείσδυσης ή για τα στοιχεία που αφορούν τη διείσδυση από τρίτα κράτη στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το να τηρούνται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου αλλά τι κάνουμε πρέπει να διαρωτηθούμε, τι είδους νομοθεσία είναι αυτή. Αυτή είναι μια νομοθεσία η οποία αφορά τις δημόσιε συμβάσει. Δεν βλέπω κανένα λόγο να Υπάρχει μια επιπλέον λοιπόν οδηγία ή ένα νομοθέτημα το οποίο ήδη έχει καλυφθεί από προηγούμενα νομοθετήματα. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία ήδη ισχύουν. Είναι τελείως περιττό το νομοθέτημα. Μας καλύπτει απόλυτα η ε, γενική οδηγία γιατί και, στην, και αυτή προβλέπει την αυστηρή τήρηση των εργασιακών συνθήκων για οποιονδήποτε να λαμβάνει συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δημόσια έργα. Ευχαριστώ κύριο Σφάπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, είχα ήδη το στο παρελθόν την ευκαιρία να συζητήσω το θέμα αυτό με τον εξαίρετο και αγαπητό συνάδελφο κύριο Μπαλτασάρε. Ξέρω ότι και εσείς ε, κύριε ε, ε, πρόεδρης ως Ιταλός Ευρωβουλευτής όπως ε, και ο κύριος Παλτασάρε, ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για μια θετική ανάπτυξη στην Ευρώπη ολόκληρη και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές εμπειρίες ανάλογα με τα κράτη-μέλη και την εθνική καταγωγή αλλά και τις περιφέρειες ακόμα από τις οποίες προέρχεται ο κάθε βουλευτής. Κανείς κανείς, ούτε καν οι Γερμανοί δεν πρέπει να διαπράξει το σφάλμα, να θεωρήσει ότι τα πράγματα ισχύουν παντού όπως τα ξέρει στο σπίτι του και στην πατρίδα του. Αλλά αυτό είναι το σφάλμα το οποίο νομίζω ε, διαπράττουν οι Ιταλοί συνάδελφοι. Διότι όντως υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ευρώπη οι οποίες για λόγους που θα πρέπει να διερευνήσουμε έτσι περαιτέρω έχουν καλύτερη ε, δυνατότητα, μεγαλύτερη δυνατότητα από ότι κάποιες άλλες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τον ανταγωνισμό. Παράδειγμα, στην Κίνα οι καλές ιταλικές μάρκες για κοστούμια έχουν εξαιρετική φήμη. Και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι εν γέννη θα κινδυνεύσουν, ε, η ιδέα ότι μπορεί να κινδυνεύσουν όλα τα ιταλικά προϊόντα σε περίπτωση που εισαχθεί αυτό το νομοθέτημα είναι σφαλμένη. Αντίστοιχα μπορεί κάποια ο κλάδος της γερμανικής βιομηχανίας να προβάλλει επιχειρήματα αντίστοιχα με αυτά του κυρίου Μπαλτασάρη για λόγους δικούς του. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε σε μέλημα το συμφέρον του πολίτη, του καταναλωτή και να επιτρέψουμε όσο το δυνατόν την αξιοποίηση των ευκαιριών που μας, που μας δίνει η παγκοσμιοποίηση και όχι να κλείσουμε τις πόρτες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε όπως, ε, όπως λένε οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ Μπαλτασάρα. Ευχαριστώ πολύ Προέδρε, δεν θέλω να καταχραστώ της ε, υπομονή σας και ευχαριστώ πολύ Ανδρέας για την κατανόηση για τους Ιταλούς συναδέλφους που επιδεικνύεις, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν προσπαθώ εδώ να περασπιστώ κανέναν, θέλω απλώς να εξηγήσω στην κυρία Βάιλερ ότι δεν μιλάμε για εξαγωγές, μιλούμε για συγκεκριμένο τομέα, δημόσιες συμβάσεις και θέλω να εξηγήσω ξεκάθαρα μια και πάντα έρχεται αυτή η αντιπαράθεση Γερμανοί εναντίον Ιταλών και το καθεστή. Μιλούμε για την Ευρώπη. Η χώρα μου δισεκατομμύρια ευρώ εξάγει όχι μόνο σε κοστούμια και σε κρασιά, αλλά και σε μηχανήματα, σε εργαλειομηχανές, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αυτοκίνητα. Δεν πουλάμε μόνο κοστούμια και γραβάτες και κρασιά. Αλλά εδώ το θέμα μας δεν είναι αυτό, είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρώσετε το συλλογισμό σας. Αφού δεν το πράξετε όμως θα το κάνω εγώ. Πώς μπορούμε λοιπόν να πωλήσουμε αν δεν ορίσουμε κανόνες στις δικές μας τις αγορές. Διότι εάν το κάνουμε αυτό μπορεί οι χώρες για τις οποίες, προς τις οποίες εξάγουμε να ενοχληθούν από τους κανόνες που επιβάλλουμε για τις δημόσιες συμβάσεις της χώρας μας. Αυτό θέλετε να πείτε βασικά κυρία Βάιλερ και τελικά να μας κλείσουν το δρόμο στις εξαγωγές. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για εξαγωγέ. Εδώ μιλάμε για δημόσιε συμβάσει. Εδώ μιλάμε για σιδηροδρόμου. Όταν πάει μια γερμανική εταιρεία στην Κίνα να χτίσει έναν αυτοκινητόδρομο, ξέρει πολύ καλά τι θα τη στήσουν οι Κινέζοι. Όταν έρθουν όμω οι Κινέζοι να χτίσουν εδώ δρόμο, δεν θα του στήσουμε το ίδιο πράγμα. Δεν καταλαβαίνω πια τι λέτε. Η βασική αρχή είναι η αμοιβαιότητα. Είναι ένα ζήτημα αξιοπρέπειας, είναι ένα ζήτημα ισχύω που δεν μετράται μόνο σε δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει τη δική του αυτόνομη αξία. Και διαφορετικά, αν δεν το κάνουμε, πολύ φοβάμαι ότι ε, μα πουλάνε το σχοινί με το οποίο θα μα κρεμάσουν κιόλα. Θα κρεμαστούμε μόνοι μα. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Νομίζω ότι η ανάλυση του κυρίου Μπαλταζάρη για την ε, τρέχουσα κατάσταση βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όταν εξετάζαμε την κατάθεση αυτής της πρότασης. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ε, πλέον αντιμετωπίζουμε σοβαρές δυσκολίες. Ακόμα και όταν έχουμε ενεργούς διαπραγματεύσεις με τους ε, εταίρους μας. Ε, δυσκολευόμαστε να μπούμε πραγματικά στις προμήθειες. Το ερώτημά μας είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Και ο λόγος, και είναι και ένα επιχείρημα που ακούμε πολύ συχνά από τους εμπορικούς μας εταίρους, Μα λένε λοιπόν ότι καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις σα σας ε, αναφέρουν προβλήματα πρόσβασης, όμως... Οι δικέ μα επιχειρήσει δεν έρχονται να μα χτυπήσουν την πόρτα και να μα ζητήσουν καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Επομένω, εφόσον πλέον είναι ικανοποιημένε οι εταιρείε από του όρου πρόσβαση, γιατί να πούμε στη διαπραγματεύσει με εσά. Είναι πολύ μικρό το κίνητρο λοιπόν για τη διαπραγμάτευση και αυτό, αυτή τη δυναμική προσπαθήσαμε να αλλάξουμε ε, για να μην μπούμε στο άλλο άκρο του, το να κλείσουμε λέει, την αγορά. Θέλουμε λοιπόν μια, ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τους όρους πρόσβαση στην αγορά και αυτό θέλω να απαντήσω και σε όσους προβληματίζονται ιδιαίτερα να μην αναφερόμαστε σε προβλήματα που δεν υπάρχουν. Γιατί οι επιχειρήσεις μας έχουν ε, μεγάλες επιτυχίες σε κάποιους ε, τομείς. Η πρόταση αυτή αφορά μόνο χώρες όπου υπάρχουν ε, συστηματικά προβλήματα διακρίσεων με ορισμένες επιχειρήσεις. Ούτε καν ε, είναι αυτό το πνεύμα του κανονισμού να δημιουργήσουμε πρόβλημα που δεν υπάρχει σήμερα. Εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης για την Ευρώπη, ε, δεν μας αφορά αυτό το εργαλείο, γιατί ούτε κλείνει τίποτα την πρώτη μέρα. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες που προβλέπονται για να ξεκινήσει διαδικασία κλεισίματος της αγοράς. Δεν συμβαίνει λοιπόν τίποτα για τα κάτω από τα 5 εκατομμύρια. Έχουμε κάνει την τεράστια υποχώρηση και λέμε ότι αυτές οι αγορές θα μείνουν ανοιχτές ε, ε, πάση θυσία. Επομένως και η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης... Ε, α, να επανέλθω τώρα σε κάτι που συνδέεται με αυτή τη συζήτηση για το ποιοι είναι πραγματικά οι όροι πρόσβασης στην Ευρώπη. Αν δείτε, αυτό αναφέραμε και στην αξιολόγηση αντικτύπου που μας ζήτησε το Κοινοβούλιο, είναι ότι αν δούμε πώς οι ξένες επιχειρήσεις παίρνουν πρόσβαση στην Ευρώπη, πρέπει να δούμε και τις ξένες θηγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη. Και θα δείτε ότι αυτές έχουν περίπου 40% της αγοράς προμηθειών στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να είναι πολύ θετικό γιατί έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό και κανένα δεν αντιτίθεται στον ανταγωνισμό επί της αρχής. Όμως όταν βλέπουμε τέσσερι χώρε να κλείνουν προοδευτικά σταδιακά τι αγορέ τους, είχαμε πρόσφατα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ε, για αυξανόμενα προβλήματα στην Κίνα, άλλες χώρες ε, στη διάρκεια των ετών, ακόμα και χώρες που δεν, παραδοσιακά δεν έχουν προβλήματα στον εμπορικό τομέα, μετά από την κρίση πήραν, έκαναν βήματα που οδηγούν σε κλείσιμο της αγοράς. Εμείς ε, καλύτερα να πούμε ότι πρέπει να προετοιμαστούμε, να εξοπλιστούμε για να έχουμε τα κατάλληλα επιχειρήματα όταν διαπραγματευτούμε με αυτούς τους εταίρους να του δώσουμε και κίνητρο να μπουν στη διαπραγμάτευση για να μην παίρνουν ω δεδομένη την ανοιχτή πρόσβαση. Και αυτό είναι ο στόχο τη ε, πρόταση. Βεβαίω και μπορείτε να απολαύετε του δικαιώματο, αλλά δεν είναι δεδομένο. Και αν ε, ξεκινήσετε τι διακρίσει ε, κατά των επιχειρήσεών μα, έχουμε κι εμεί μέσα και εργαλεία για να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Όμως δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον κάποιου που δεν είναι κάνει διακρίσεις. δεν είναι ένα μέσο το οποίο θα αφορά τους πάντες. Αντιθέτως, το έχουμε προετοιμάσει πολύ προσεκτικά για να αφορά χώρες που ε, κάνουν συστηματικά διακρίσεις, ιδίως ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Βεβαίως, αυτό είναι στα χέρια του εισηγητή Πρέπει να δούμε πώ ε, θα χειριστεί τι ε, διάφορε τροπολογίε που έχουν κατατεθεί και βεβαίω είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί του. Όμω ε, στην βασική ανάλυση τη τρέχουσα κατάσταση υπάρχει πρόβλημα. Εμεί προτείνουμε μια λύση, μπορούμε να το εξετάσουμε το θέμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μα και η μεγαλύτερη επιφύλαξη είναι ότι σε κάποια σημεία δεν αναγνωρίζουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει και επιδεινώνεται. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Αλλά βεβαίω θέλουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και του υπολείπου σε αυτό. Υπάρχουν πολύ καλέ ιδέε έτσι κι αλλιώ, τι οποίε μπορούμε να επεξεργαστούμε. Θα μείνω εδώ προ το παρόν. Να μην υψέλθω σε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Φρανκ. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω στους Ιταλούς ε, συναδέλφους ότι κατά τη γνώμη μου, ναι πράγματι έχετε δίκιο, ισχύουν τα όσα λέτε, αλλά δεν αφορούν τη σημερινή συζήτηση. Για μένα τουλάχιστον. Προβλήματα που ενδεχομένως να έχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους σε, άλλα, σε άλλες χώρες του κόσμου, αφορούν ε, τις τιμές ή άλλους παράγοντες, γιατί απλώς δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Σίγουρα αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Όμως, κατά τα λοιπά, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι, οι Βραζελιάνοι, οι Ρώσοι, εφόσον αποφασίζουν να θεσπίσουν ε, τέτοιες πολιτικές του buy local, buy national ε, πρόκειται για έθνη, για κράτη και γι' αυτό μπορούν να πάρουν τέτοιες αποφάσεις. Εμείς δεν είμαστε ένα ενιαίο κράτος, επομένω δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια απόφαση. Ουσιαστικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που ε, μεριμνούν την υπεράσπιση των συμφερόντων του. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας Ιταλό, ένα Γερμανό, ένα Βρετανό πάντα ε, φροντίζει να έχει μια προβολή στην Κίνα, ακόμα και αν αυτό έρχεται σε βάρος ε, του Ισπανού ή του Σουηδού. Αλλά αυτή είναι μια εγγενής ε, αντίφαση της Ευρώπης. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ή να λύσει την, επιλύσει το πρόβλημα, γιατί το σχέδιο γνωμοδότησης δεν αφορά αυτό το θέμα. Λοιπόν, Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνάφεια ή μη ενός τέτοιου εργαλείου, το καλύτερο θα ήταν να πούμε ότι δεν θα επιλύσουμε ε, το πρόβλημα αν δεν αναγνωρίσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και άλλοι. Σε διμερείς συμφωνίες που μπορούν να πάρουν άλλη μορφή στο μέλλον και με πιο σταθερή θέση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο διεθνές προσκήνιο. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να επιλύσουμε το πρόβλημά μας. Το σχέδιο κανονισμού δεν θα τα καταφέρει. Όταν ξεκίνησε, αν θέλετε η πρώτες κανονισμού, υπήρχε ε, μια ε, μικρή εκδήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Μάρκε Χάμπερ και ανέφερε ένα αριθμητικό στοιχείο. Είπε ότι περίπου 30 οντότητες ε, θα αφορά αυτό το κείμενο. Επομένω, η λύση εδώ πέρα δεν είναι πανάκια, συμφωνούμε. Όμως, το κείμενο έχει τεθεί επιτάπητος. Προσπαθήσαμε να το διατηρήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι συμφωνίε δημοσίων προμηθειών, θα πρέπει αλλιώ ε, να γίνονται διαπραγματεύσει στο μέλλον. Και αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ε, ουσιαστικά εδώ πέρα γνωμοδότηση κάνουμε, επομένως θα διατηρήσω την ηρεμία μου. Καθώς ε, οι συνάδελφοι δεν είναι τόσο μεγάλοι υποστηρικτέ ε, του κειμένου, ούτε θα, επομένως δεν θα επιληθούν όλα τα εμπόδια πρόσβασης στις δημοσίες προμήθειες. Ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε αργότερα σε αυτό το θέμα. Και θέλω να καθησυχάσω τον Γερμανό συνάδελφο για να πω ότι δεν υπάρχει γερμανική, ή ιταλική άποψη ότι υπάρχει δηλαδή αντιπαλότητα μεταξύ μας. Όχι. Δεν θα μιλούσα καν αν ήξερα ότι θα δημιουργηθεί σύγχυση. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα περάσουμε στο τελευταίο σημείο. Ε, έκθεση Κοράτσα Βίλντ για την απάτη ε, στην ε, αλυσίδα τροφίμων. Θα μιλήσω αγγλικά. Συνάδελφοι, αυτή η γνωμοδότηση ε, αφορά το πώς θα οικοδομηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη στην ε, αγορά τροφίμων. Μετά από όλο το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, πολλοί πολίτες μας ανησυχούν ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα από χώρες που έρχονται από, από κρέας που έρχεται από τρίτες χώρες. Ε, και θεωρούν ότι δεν μπορούν να εμπιστεύονται πλέον ε, το, το φαγητό που τρώνε και θεωρώ ότι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι τρώνε. Κύριε Πρόεδρε, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει νέο νομοθέτημα ή προστιθέμενη νομοθεσία, όμως ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού χρειαζόμαστε για να είμαστε σίγουροι ότι ε, με τους κανόνες που έχουμε, έχουμε τα, τα υψηλότερα ε, διατροφικά πρότυπα στον κόσμο, ότι αυτά τα πρότυπα λοιπόν εφαρμόζονται με τον κατάλληλο τρόπο. Λοιπόν, στρέφουμε προς την Επιτροπή. Το σύστημα ε, κοινοποίηση, απαγρύπνηση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσε πολύ καλά. Ο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών λειτουργήσε πολύ καλά και η Επιτροπή κατάφερε πολύ γρήγορα μετά από τεράστιο όγκο ε, τεστ DNA να καθησυχάσει τους ε, πολίτες ε, το ότι δεν πρόκειτο για κρίση επιστημικής ασφάλειας αλλά σήμανσης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί οι παραπλανητικέ πληροφορίε και τα ψεύδη είναι το πρόβλημα, όχι το κρέας αλόγου. Είναι σημαντικό να το γνωρίζει ο πολίτη. Ε, τι σημαίνει αυτό, τι περιέχει το τρόφιμο που αγοράζει και να κάνει ε, ε, μια τέτοια επιλογή. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, θα πρέπει να είναι πιο σαφής ο ορισμός της απάτης στο γενικό δίκαιο τροφίμων και ε, στην αντίστοιχη οδηγία. Προ το παρόν, οι παραπλανητικέ πληροφορίε απαιτούνται μόνο όταν πρόκειται για κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει να καταστεί σαφέ και να επεκταθεί και στι περιπτώσει ε, παραπλανητικών πρακτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, σήμανση προέλευσης, τα έχουμε συζητήσει αυτά και στο παρελθόν, κατά την υιοθέτηση νομοθεσίας για τη σήμανση και έχουμε συμπεριλάβει υποχρεωτική ε, σήμανση για κάθε είδους κρέατος. Και περιμένω να δω και τις ε, εκτελεστικές πράξεις για να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, για να μην ε, δημιουργήσουμε περισσότερα κόστη και διαδικασίες για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς. Και αυτό θα έρθει μέσα στον επόμενο χρόνο. Όμως χρειάζομαστε καλύτερη χναλισιμότητα, διαφάνεια σε μια αλυσίδα που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και ε, αφορά πολλές χώρες. Επομένω, ε, είναι πολύ θετική η εξολόγηση αντικτύπου ε, της Επιτροπής για την εθελοντική σήμανση κρέατος. Και θεωρώ ότι θα ήταν καλό να περάσουμε σε μια τέτοια σήμανση. Δεν θα πρέπει να μπούμε στην συζήτηση, δηλαδή αν πρέπει να υπάρχει σήμανση για το ε, κρέας όταν ε, πρόκειται για συστατικό, όπως αυτή η κουβέντα που είχε γίνει με τα λαζάνια. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό ή ε, ότι θα έχει προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή να έχουμε σήμανση για κάθε ξεχωριστό συστατικό των τροφίμων. Γιατί τελικά θα βγουν από την αγορά οι μικροί παραγωγοί. Και βεβαίω μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό περαιτέρω. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι θα διαφωνήσουν. Άλλο σημείο που είναι σημαντικό για μένα είναι οι κυρώσει. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώ ε, ανέμακτες αυτές οι κυρώσει Δεν μπορούμε να, δούμε τη δυνατότητα να υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος ε, για, τον, ε, για την επιχείρηση, ώστε να είναι διατεθειμένη να αναλάβει τον ε, κίνδυνο. Ε, πρέπει να έχουμε λοιπόν κυρώσει που να αποτρέπουν, να αποθαρρύνουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τι επιχειρήσει από το να ακολουθήσουν παραπλανητικές μεθόδους. Αυτό μπορεί να εξεταστεί σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας μέσω της επιβολής, της καλύτερης επιβολής και εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των αρχών κρατών μελών. Στα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι Έχουμε πολύ λίγες υποθέσεις απάτης ε, στην ε, αλυσίδα τροφίμων που οδηγεί ε, στην νομική δράση. Και θα ήταν καλύτερο να ενθαρρύνουμε ε, τέτοιου είδους ε, υποθέσεις, να υπάρχει κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, να είμαστε σίγουροι ότι αυτό ε, εξετάζεται πολύ σοβαρά. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ακούσω τους συναδέλφους, τους κοιόδης και να σας υπενθυμίσω ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάσταση των προλογιών είναι αύριο Σίγουρα θέλω να εξετάσω και το ζήτημα των ιδιωτικών ετικετών, γιατί τμήμα του σκανδάλου ε, που αφορά το κρέας αλόγου αφορούσε τις ιδιωτικές ετικέτες. Δεν χρειάζεται να δαιμονοποιήσουμε βεβαίως κανέναν. Από επιστημονική σκοπιά θα πρέπει να δούμε αν οι ιδιωτικέ ετικέτες δίνουν τις ε, ε, σωστές πληροφορίες, τη διαφάνεια και την ελεύθερη επιλογή για τους καταναλωτές που θέλουμε να διασφαλίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η διορία κατάθεση τροπολογιών λίγη το μεσημέρι αύριο, 27 Σεπτεμβρίου, όπως είπατε κι εσείς. Και αφού θέλει ο εισηγητής να ακούσει τις απόψεις των συναδέλφων του, ορίστε η κυρία Βάιλερ των Σοσιαλιστών. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Καλό θα ήταν ίσως η διορία κατάθεση τροπολογιών να λύγει αύριο, αν και είναι σύντομο το χρονικό διάστημα και οι περισσότεροι θα είναι, δεν θα είναι πια εδώ αύριο, αλλά είναι επίσης καλό να γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος εδώ και χρόνια ασχολείται με το θέμα αυτό της απαραίτητης σήμανσης. Ήθελα και εγώ να καταθέσω τροπολογίες, αλλά το αφήνω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εδώ πρόκειται για θέμα υγείας, όπως ξέρετε. Και δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια, χρειάζονται συγκεκριμένοι κανόνες. Πρόκειται και για θέμα αναπτυξιακής βοήθειας, πρόκειται για θέμα δυσπιστίας των καταναλωτών και καταναλωτριών και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι οι καταναλωτές σε τέτοια θέματα. στα υγειονομικά και διατροφικά σκάνδαλα δηλαδή. Χρειάζεται λοιπόν απαραίτητο εδώ διαπάνεια. Όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και για τους παραγωγούς και για τους απατεώνες που πρέπει να αποθαρρυνθούν και με αυτή την οδηγία της διαφανείας θα διευκολυνθούν, θα βελτιωθούν τα πράγματα αλλά ούτε η διαφάνεια αρκεί. Σε περιπτώσεις απατών η διαφάνεια εδώ από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα και ούτε η αυτορύθμιση. Πάντοτε υπάρχουν τα μαύρα πρόβατα που είναι και αρκετά πολύ άριθμα και η αυτορύθμιση είπα δεν αρκεί και δεν υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι. Και νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τη διαμεθοριακή διάσταση παραπάνω από ό,τι το κάνει το αρχικό κείμενο. Από την Ιρλανδία ως τη Σλοβαϊνία Σλοβακία, μερικά προϊόντα περνάνε τα σύνορα και του αλλάζει η σήμανσή τους και μερικές φορές επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης. Είμαστε σε μια, βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα και αυτό διευκολύνει κάπως τις απάτες. Da sind ja sogar die Regierungschefs schon ein bisschen weiter. Die haben nämlich im Sommer beschlossen. Το είπαν και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ότι Χρειάζονται νόμοι, νομοθετήματα κατά της κερδοσκοπίας, αλλά και σε αυτό το θέμα των τροφίμων χρειάζεται. Για να βελτιωθεί η κατάσταση και στις τρίτες χώρες και στις ενουσιακές, στις αναπτυσσόμενες και πρέπει να υπάρξει επίσης βελτίωση για τα αγροκτήματα, για τους δήμους και κοινότητες, για πολλά πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν θετικά στοιχεία, αλλά πρέπει να βάλουμε τη διαφάνεια μπροστά μπροστά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Α, ευχαριστώ πρόεδρε. Υπήρξαν μεγάλα σκάνδαλα, ιδίως με το κρέας. Υπήρξε η γρήπη των πτηνών, όπως θα θυμάστε και άλλες τέτοιες κρίσεις. Του... Μπορεί κανείς να πει λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, σκανδαλίστηκαν και πολύ δοκιμάστηκαν. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για την πρόταση που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή μια σαφέστερη σήμανση των τροφίμων θα μπορούσαμε όμως ίσως να τονίσουμε περισσότερο το θέμα των κυρώσεων. που πολλοί το θεωρούν λεπτομέρεια. Δεν γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι και οι κυρώσεις είναι πολύ χαμηλές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι πρέπει να είναι βαρύτερες και πιο αποτρεπτικές οι κυρώσεις. Επίσης, να κυρώνεται και η μη δήλωση. Να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Σε εθελοντική σήμανση γιατί όχι, αλλά για να υπάρξει εμπιστοσύνη χρειάζονται κυρώσεις. Ε, μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ συζητιέται αυτή τη στιγμή και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ίδια η έλεγχη παντού. Το βλέπουμε αυτό. Το γάλα σε σκόνη είναι τεράστιο πρόβλημα στην Κίνα. Το 8 ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Γιατί... Και μετά έχουμε τις φράουλες. Και έτσι νομίζω ότι θα ήταν καλό να, κάνουμε, να δώσουμε έμφαση στον έλεγχο των εισαγωγών για να διατηρήσουμε, να διαφυλάξουμε την ποιότητα στις αγορές μας. Άρα ναι, πρέπει να έχουμε την ένδειξη προελεύσεως, αλλά ταυτόχρονα και όταν έχουμε διμερείς συμφωνίες να κοιτάμε και τα θέματα αυτά. Μπορεί λοιπόν να χαρακτηρίζομαι ως ε, ε, ακραίος φιλελεύθερος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια αγορά με, με, καλά, με, με καλούς ελέγχους και βεβαίως συμπρολέψεις. Ευχαριστώ πολύ, δεν είναι έχεις της κανένας άλλο το λόγο. Η κυρία Ρούιλε. Πρόεδρε, όλο με αγνοείται, αλλά θα ζήσω. Ίσως νομίζουν αυτομάτως όλοι ότι ανήκουμε σοσιαλιστές, αλλά θέλω να κατασ... Απόλυτα σαφές ότι δεν ισχύει αυτός ο επινιγμός. Όχι, λέει ο κύριο Κοφεράτη, το έχω καταλάβει εδώ και καιρό. Μέσα περιπτώσει, για την διαφάνεια, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι ε, χρειάζεται ε, να υπάρξει αυτή η πρόταση για τον έλεγχο για την ε, επαλήθευση δεν χρειάζεται περαιτέρω αλλαγή. Στα 5, 6, 7 μπορούμε να σας υποστηρίξουμε, αλλά στο 1 και στο 3 δεν μπορούμε να σας ακολουθήσουμε, διότι θεωρούμε ότι η εθελοντική ε, σήμανση ανήκει πια σε παροχημένες εποχές. Χρειαζόμαστε πλέον περισσότερη διαφάνεια, πολύ περισσότερη διαφάνεια, την οποία η ε, εκούσια σήμανση δεν καλύπτει. Ναι. Οι φράουλες από την Κίνα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Θέλω να ξέρω τι τρώνα τα παιδιά μου. Δεν μπορεί λοιπόν στα τρόφιμα να μην έχουμε σήμανση προέλευσης. Αυτό μας προξενεί πάρα πολλά προβλήματα. Και για το κρέας ασφαλώς. Δεν μπορεί δηλαδή να ε, παίρνει κανείς προϊόντα από 6, 7, 8 διαφορετικά κράτη και από, αυτά τα προϊόντα να φτιάχνει μια πίτσα. Πρέπει να, από το ίδιο κράτος να είναι όλα από, το, από μια χώρα να πάρει τα λουκάνικα, να πάρει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί λοιπόν ναι, ναι. κάθε φορά να έχουμε από διαφορετικά προϊόντα και να μπαίνουν όλα πάνω σε μία πίτσα. Μόνο να παραπλανήσουμε τον καταναλωτή μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Κάτι το οποίο προσπαθούμε να αποφύγουμε προφανώς. Δυστυχώς όμως ε, δεν ε, προλάβαμε, να, δεν προλάβαμε τις, ε, τις προθεσμίες για τις τροπολογίες και γι' αυτό θα χρειαστεί να απορρίψουμε τροπολογία σας και τα σημεία, την έκθεση σας και τα σημεία 3, 4, 5 μας αρέσουν πάρα πολύ. Η κυρία Κάρμεν Γκράου για την Επιτροπή. με συγχωρείτε, κύριος Μπίλαν. Ο κύριος Μπίλον. Ο οποίος δεν πιστεύω να με κατηγορήσει και αυτός ότι τον ε, παίρνω για σοσιαλιστή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι, δεν ανήκω στους σοσιαλιστές, ούτε εγώ. Χρόνο δεν έχουμε, το ξέρω. Θυμόμαστε όλοι το σκάνδαλο με το κρέας αλόγων και την κυκλοφορία του στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Η πρόταση της κυρίας Κοράτσα είναι καλή, πράγματι, και κυρίως τα σημεία που αφορούν την εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο των διατάξεων για τα τρόφιμα που περιέχουν κρέας ή προϊόντα κρέατος και εγώ υποστηρίζω την καλύτερη ανιχνευσιμότητα ή ίχνη λαυσιμότητα και υλοποίηση. Περισσότερο συντονισμό επίσης θα προτείνω μεταξύ των εθνικών αρχών ε, ε, επιτήρησης της ποιότητας των τροφίμων ή της δημόσιας υγείας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε προβλήματα και να έχουμε πιο έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων, των όποιων προβλημάτων. Καλύτερη λοιπόν προσ... περισσότερη προσπάθεια για συντονισμό και ε, οργάνωση. Επίσης, όταν διαβάζει κανείς ένα κατάλογο συστατικών σε ένα προϊόν, καταλαβαίνει ο καταναλωτής πραγματικά τι είδους είναι αυτά τα συστατικά και πόσο μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του. Γιατί εδώ εγώ δεν θα έλεγα ότι ο κίνδυνος είναι τόσο η απάτη ως προς την αλυσίδα της ε, προμήθειας, αλλά η κατανόηση πλευρά του καταναλωτή των συνεπειών ενός ε, προϊόντος. Ευχαριστώ τώρα η κυρία Γκράου. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα μιλήσω ε, αγγλικά. Λέει ο ομιλήτρια και μιλάει ιταλικά. Ναι, για τα σκάνδαλα της απάτης. Πράγματι, δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ ένας ορισμός της απάτης. Λέει μόνο απατηλές πρακτικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε πραταβουλίες για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που συνεχώς αυξάνεται ιδιαίτερα διότι άλλος πυλών της διατροφικής αλυσίδας είναι ακριβώς η υποχρέωση των χωρών μελών να διασφαλίζουν και να επαληθεύουν το σεβασμό της διατροφικής αλυσίδας από όλους τους παράγοντες και ανασέβονται όλοι, όλες τις υποχρεώσεις τους από την παραγωγή τη διανομή. Άρα είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να ταυτίζουν και τις ηθελημένες παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη διατροφική αλυσίδα. Αυτό είναι που δεν έγινε με το σκάνδαλο του αλογίσιου κρέατος. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα σύστημα γρήγορης ταύτισης του προβλήματος και του μεγέθους του διαμεθοριακός. Γιατί πολλοί μιλάνε για εναρμονισμένο ορισμό του τι είναι διατροφική απάτη, αλλά το πρόβλημα μπορεί να λυθεί και χωρίς αυτή την εναρμόνιση. Όλες οι χώρες μέλη ξέρουν περίπου τι είναι απάτη και προβλέπουν κυρώσεις. Τι κάνει λοιπόν η Κομισιόν. Υπάρχει μια πρόταση του περασμένου Μαΐου με στόχο συγκεκριμένα την ενδυνάμωση της εργαλειοθήκης μας, τη toolkit όπως λέμε, που να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να σέβονται την νομοθεσία. Ιδίως ένα νέο στοιχείο είναι ότι πρέπει τα κράτη-μέλη εθνικά σχέδιά τους να έχουν ένα συγκεκριμένο τμήμα που να μιλάει για ευνηδίους απροειδοποίητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν υπάρχουν οι θελημένες παραβιάσεις. Τώρα λοιπόν γνωρίζουν την υποχρέωση αυτή τα κράτη-μέλη και πρέπει να τα σέβονται όλα αυτά. Και στο εξής και συγκεκριμένα τις απάτες. Δεύτερη αλλαγή αφορά τις κυρώσεις που αναφέραν πολύ. Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στην τυποποιημένη ρήτρα που έχουμε σε όλες μας τις νομοθεσίες που απαιτεί από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν οικονομικές κυρώσεις που είναι η κοινότερο είδος κυρώσεων, πρόστιμα δηλαδή, σε επίπεδο που να αποζημιώνει. Όταν δηλαδή καθοριστεί το επίπεδο πρέπει να καθοριστεί μετά τι όφελος θα είχε ο απατεών για να καθοριστεί έτσι αναλόγως και το πρόστιμο. Άλλα που κάνει η Κομισιόν εκτός από τη νομοθετική πρόταση που σας ανέφερα είναι ότι κάνει ένα stepping up της ε, αντιαπατεωνικής μας δυνατότητας Με τη δημιουργία ενός δικτύου για τις τροφικές απατεωνίες. Δημιουργήθηκε λοιπόν το δίκτυο συνεδρίασαν μία φορά τα μέλη του και θα ξανασυνεδριάσουν με στόχο να αυξηθεί η δυνατότητα του συστήματος να ανοιχνεύει, να προβλέπει τις απάτες και να αντιδρά με γενικότερο πλαίσιο την νομοθεσία που ισχύει για όλους τους επίσημους ελέγχους και τη διοικητική βοήθεια και συνεργασία μεταξύ χωρών μελών σε περίπτωση διαμεθοριακών παραβιάσεων της νομοθεσίας για την τροφική αλυσίδα. Δηλαδή έχουν την υποχρέωση τα κράτη-μέρη να αλληλοβοηθούνται σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου. Τώρα καθορίζουμε ένα πλαίσιο όπου να μπορεί να υπάρξει πιο αποτελεσματική τέτοια συνεργασία όποτε είναι η θελημένη και με οικονομικό κίνητρο η παράβαση και μια από τις προτεραιότητες της ομάδας αυτής εκτός από τη δημιουργία του επίσημου μηχανισμού είναι και η βελτίωση των, της τεχνογνωσίας για αυτό το θέμα. Μερικοί είπαν και είναι πράγματι πολύ σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής μας ότι υπάρχει και η ανάγκη να αυξηθεί συνεργασία μεταξύ τροφικών εποπτών για να διασφαλίζεται ότι η τεχνογνωσία που στοχεύει στην καταπολέμηση των απατών θα είναι πραγματική. Συνεργασία λοιπόν και λοιπά. Τουλάχιστον η μεγάλη προτεραιότητά μας αυτή είναι και βέβαια γίνονται πολλά ακόμη και αν δεν έχουμε ακόμη επίσημο ορισμό της απάτης. Ε, ίσως να σταματήσω εδώ, ίσως μήπως θέλουν οι συνάδελφοί μου να προσθέσουν τίποτε για τις σημάνσεις. Μα ναι, ναι, ναι. Τι προβλέπετε για την σήμανση υποχρεωτική, εθελοντική κλπ. Πρώτον, είμαστε on track με, για τους κανόνες για την υποχρεωτική σήμανση για το αμεταποίητο κρέας και εγκαίρως θα σας γνωστοποιήσουμε και επίσης για τους κανονιστικές διατάξεις για την εθελοντική σήμανση. Όταν για τι προβλέπετε για την υποχρεωτική σήμανση του κρέατος ως στοιχείου. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε μια πλήρη αξιολόγηση, αλλά η έκθεσή μας είναι in the pipeline όπως λέμε. Θα παίρνει υπόψη της τις επιπτώσεις της μικρομεσαίες επιχειρήσης, καταναλωτές και τα λοιπά. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, εμείς σας ευχαριστούμε. Συγητή, Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις σημαντικότατες συμβολές τους στη συζήτηση και θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε οι πολιτικές ομάδες για να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το είπε και η Κομισιόν, πολλά γίνονται και χρειάζεται εδώ μια ισορροπημένη προσέγγιση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εδώ κοινωνιοδημοκράτες, αλλά θα ήθελα να πω και σε εκείνους και στους πράσινους ότι θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο επικοδομητικότεροι για να δούμε... Εκτός από κύριε από Ποια είναι τα θετικά στοιχεία και τι άλλο προτείνουμε. Η γνωμοδότηση δεν είναι βίβλος. Έχει πολύ μικρές δυνατότητες ε, και από την ανάλυση που έχουμε στα χέρια μας βλέπουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια για περισσότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Άρα και καλύτερος ορισμός. Δεν είμαι κατά της σήμανσης προέλευσης, είμαι από εκείνους που το ζητούσαν για όλα τα κρέατα στην πολιτική μου ομάδα. Λέω όμως ότι αν θέλουμε πράγματι να στηρίξουμε την αγορά και να δοθούν ίσες ευκαιρίες και στους καταναλωτές και στους μικρομεσαίους ε, παραγωγούς, η απάντηση δεν είναι με νομοθετικές διευθετήσεις, γιατί η υπερβολική νομοθεσία δημιουργεί μεγαλύτερα διοικητικά βάρη και άχθη σε εκείνους ακριβώς που πρέπει να στηρίξουμε. Πρέπει να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των καταναλωτών με τρόπο όμως που να τους ωφελεί και επίσης να προσπαθήσουμε να μην βγάλουμε από την αγορά εκείνους ακριβώς τους παράγοντες που θέλουμε να βοηθήσουμε. Και θα ήθελα η κυρία Ρούλα να αναθεωρήσει. Ξέρω ότι είναι λίγος ο χρόνος, αλλά είναι σημαντικό να προχωρήσουμε, να βρούμε απαντήσεις για αυτό το θέμα που δημιουργεί τόσες αντιδράσεις και προς τους καταναλωτές και προς τις εταιρείες. Η γνωμοδότηση δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου. Μη μου λέτε λοιπόν ότι θα καταψηφίσω γιατί δεν προλαβαίνω τις τροπολογίες αύριο. Εγώ δεν μπορώ να πω στους ψηφοφόρους μου ότι δεν ψήφισα ή καταψήφισα γιατί δεν πρόλαβα να γράψω τροπολογίες δεν είναι θέμα ασφαλείας των τροφίμων, είναι θέμα καταναλωτικό. Ε, καταναλωτικό. Δεν πρέπει λοιπόν να αρνηθούμε τις ίδιες μας τις ευθύνες. Και πιο συγκεκριμένα κύριε Πρόεδρε θέλω επίσης να απαντήσω στο συνάδελφό μου από την Επιτροπή ΕΛΕΦ το λέει και η γνωμοδότηση ότι ζητούμε περισσότερους και καλύτερους ελέγχους και υποχρεωτικούς μάλιστα. Με τρόπο όμως που να μην είναι απλώς τιμωρητικός, γιατί μερικές φορές υπερβολικά πολλοί έλεγχοι για μικρές εταιρείε δημιουργούν προβλήματα. Ο χρόνος είναι χρήμα για αυτές. Και να, να πανίσουν τρεις μέρες για τον έλεγχο της βλάπτει. Πρέπει λοιπόν να παίρνουμε υπόψη μας και την πραγματικότητα των μικρομεσαίων εταιριών. Πρέπει στις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις και με τα Συνωμένας Πολιτείας να τηρήσουμε σταθερή στάση. Και αυστηρότερες κυρώσεις. Αλλά βέβαια αυτά εθνικά. Εδώ περιοριζόμαστε στην ανταλλαγή εμπειριών. Δεν νομίζω ότι κυρώσεις εφαρμόζονται ενωσιακώς. Το χρονοδιάγραμμα που μας επιβάλλει η ΕΝΒΗ μας πιέζει γιατί έχουν και άλλη έκθεση και θέλουν την γνωμοδότησή μας πριν. Ευχαριστώ. Και προσβλέπω σε τροπολογίες. και στη συνεργασία των συναδέλφων και της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Γεια σας όλοι. Θα ξαναδούμε το απόγευμα. Sì, oggi pomeriggio c'è la tavola rotonda in continuazione proprio con almeno ναι, σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη στρογγυλή τράπεζα και ενδεχομένω να συνεχίσει αυτή η παρακολούθηση σε άλλη, σε άλλη συνεδρίαση. Και βεβαίως αυτό συνδέεται και με την ευαισθητική ασφάλεια, αλλά όχι μόνο.